Jest Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα την έκτακτη μας συνεδρίαση που προβλέπει ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών κατά των πειραμάτων σε ζώτα ζώα κοινή συνεδρίαση. Επιτροπή των Αναφορών, Επιτροπή Περιβάλλοντος Νόσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω πως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών θεσπίστηκε με τον κανονισμό 2000, του 2011 με τον αριθμό 211 που στόχο είχε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να διατυπώσουν τις ιδέες τους και να, ζητούν, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση πρωτοβουλίας σε θέματα αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύκολο να το λες. Αλλά η δουλειά δεν είναι καθόλου εύκολη. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι μια πρωτοβουλία απαιτείται να συλλέξει ε, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές πολιτών προερχομένων από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να εξετάσει το αίτημά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχοντας λοιπόν αυτό το γεγονός υπόψη, αυτή την προϋπόθεση υπόψη, θέλω να συγχαρώ τους ε, διοργανωτές τον κύριο Αντρέι Μένας που είναι εδώ, τον κύριο Τζάνι Ταμίνο και τον κύριο Κλωτράης που οργάνωσαν αυτή την πρωτοβουλία. Εκπροσωπούν από κοινού την οργανωτική ομάδα της πρωτοβουλίας και θα θυμάστε ίσως ότι έχουμε ξανακάνει ακροάσεις, πρόκειται για την τρίτη ακροάση στο θέμα αυτό. Μάλλον τρία διαφορετικά θέματα για να είμαι ακριβής. Οι προηγούμενε εκδόσει αφορούσαν ε, ε, το θέμα των υδάτων και προέρχονταν πάλι από πρωτοβουλία των πολιτών. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τους ειδικού μας. Τον κύριο Γκρικ πρώτα, yes. πρόεδρο της Αμερικανικής Εταιρείας Ιατρικής Προόδου. Την κυρία Μπαρέσινουσή, καθηγήτρια στο, στο Ινστιτούτο Παστέρ βραβευθήσα με το βραβείο Νόμπελ το 2008, βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Σας καλωσορίζουμε, χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ. Και την κυρία Μακάιβορ, μέλος της Ανθρώπινης Εταιρείας Διεθνούς. Όπως έλεγα λοιπόν, είναι η συνεδρίασή μας αυτή κοινή με τις Επιτροπές των Αναφορών του Περιβάλλοντος και της Βιομηχανίας. Έχουμε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να καλωσορίσω τον κύριο Ματσόλα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Αναφορών, τον κύριο Γιώργη Κατάιναν, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κύριο Καρλ Φάλκενμπεργκ, γενικό διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως για το Περιβάλλον. Πριν δώσω το λόγο στους διοργανωτές της ε, πρωτοβουλίας, θα ήθελα να μου επιτρέπετε να κάνω εγώ μια σύντομη επισκόπηση των προβλημάτων ή των ζητημάτων, ούτως πει, με το οποίο σχετίζεται η πρωτοβουλία των πολιτών. Και οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιούνται ζώα σε πειράματα, ζώντα ζώα, είναι οι πρώτη θεματολογία στην οποία θα επεκταθώ. Ε, η δε δεύτερη είναι η επιτέλεση του ρόλου που έχει προβλεφθεί από την οδηγία για τη διευκόλυνση επιστημονικής έρευνας με χρήση ζώων των ζώων. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε εάν επιτρέπει την εισαγωγή νέων επιστημονικών πρότυπων αυτή η οδηγία, όπως ισχύει ώστε να εγκαταλειφθεί η ιδέα της χρήσης ζών για την επιστημονική έρευνα. Και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση των ζών. Μια άλλη ιδέα είναι να ότι πρέπει εξάπαντας να εξασφαλίσετε και η ευημερία ή η η ευζωια των ζών. Θα πρέπει πάντω πριν παραδώσω το μικρόφωνο, να σημειώσω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με την τήρηση του χρόνου, γιατί έχουμε μόνο μέχρι τις 6,5 ε, περιθώριο για τη συνομιλία μα αυτή. Τώρα θα παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή των Αναφορών να λάβει το λόγο πρώτο. Την Αντιπρόεδρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και όπω ζητήσατε θα προσπαθήσω να μην ε, σα ε, καθυστερήσω. ω αντιπρόεδρο όμω τη Επιτροπή των Αναφορών θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη χαρά και τιμή που αισθάνομαι για την ευκαιρία που μου δίνεται να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με την ευκαιρία αυτή. Η εμπειρία μου μου λέει ότι πολλοί μπερδεύουν το ρόλο της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών και της Επιτροπής των Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία και τα δύο, με διαφορετική όμως διαδρομή. Και είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε τις διαφορές. Η η Επιτροπή μας έχει την ε, δυνατότητα να δώσει φωνή και να ενισχύσει τα επιχειρήματα κάποιου πολιτή, ακόμη και μεμονωμένου που μπορεί να υποβάλει αναφορά προς εξέταση. Σε μια περίοδο λοιπόν όπου ο πολίτης αισθάνεται αποκομμένος από τη διαδικασία ε, λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το εργαλείο της αναφοράς και της επικοινωνίας με την Επιτροπή των Αναφορών. Η, κατα... η δε εξέταση μια πρωτοβουλία πολιτών που ενδεχομένω έχει απορρίψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το επιχείρημα ότι δεν προτείνει αναθεώρηση ε, υφιστάμενης νομοθεσίας ή ε, νέα νομοθέτημα θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο ή καλύτερα τροφή εργασίας για την, Ευρωπαϊκή, για την Επιτροπή των Αναφορών. Έχουμε κάποιες, ε, κάποιους περιορισμούς ωστόσο και μέσα στην ε, περίοδο της αναθεώρησης στην οποία βρισκόμαστε τώρα, της ενδιάμεσης αναθεώρησης, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε χάρη και στην εμπειρία αυτή νέα στοιχεία. Με την πρωτοβουλία των πολιτών και τα πρώτα της χρόνια είναι ξεκάθαρη η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε τα προβλήματα ώστε να γίνει το εργαλείο αυτό στο δυνατόν πιο εύχριστο για τον πολίτη και αποτελεσματικό. Για το ενώπιον μας ζήτημα. Έχουμε δύο αναφορές για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα, ζώα και την κατάργηση σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πειραματισμοί σε ζώντα ζώα έχουν αποτελέσει πηγή πολλών συζητήσεων σε όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες είναι θέμα συναισθηματικά φορτισμένο. Γιατί έχουμε βεβαίως αντιληφθεί ότι πολλοί και εγώ ίδια έχουν ε, σαφέστατη τοποθέτηση και συγκίνονται πολύ από το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών, να συζητηθεί η θεματολογία της και να εξασφαλιστεί και η κύρωση των αποτελεσμάτων. Η οδηγία του 2010 έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο από όλα τα κράτη-μέλη. Έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2013. Στόχο είχε την επικαιροποίηση της προηγούμενης οδηγίας του 1996. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τα πειράματα σε ζώντα ζώα και γενικά τα πειράματα σε ζώα που ε, εγείρει αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή των Αναφορών θα ενημερώσει τους αναφερομένους για την έκβαση της ακρόασής μας και κυρίως για τις θέσεις που θα εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ε, τον Αντιπρόεδρο Καθάινεν. Κατά απόλυτα την τρόπο με βέβαια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κατάινεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που οργανώνετε αυτήν ε, την ε, τόσο ανοιχτή ακρόαση σήμερα για το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών κατά των πειραμάτων ζωντά Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής ε, με τη συλλογή του 1 εκατομμυρίου δηλώσεων υποστήριξης αποδεικνύει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δομή της. Είναι η τρίτη πρωτοβουλία πολιτών μετά το Right to Water και το One of Us από πέρσι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν με τη συμμετοχή τον Απρίλιο του 2012. Θέλω να υπενθυμίσω με μερικά λόγια την πρωτοβουλία των πολιτών και μετά να περάσω στο θέμα τη απόψηνή μα ακρόαση. Η Επιτροπή στι 31 Μαρτίου υιοθέτησε μια έκθεση η οποία αξιολογεί την πρώτη τριετία λειτουργία του νέου αυτού εργαλείου τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ενώ καταλήγουμε στο συμπεράσμα ότι η διαδικασία όπω προβλέπεται από τον κανονισμό για την πρωτοβουλία των πολιτών λειτουργεί ικανοποιητικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα περιθώριο ακόμη βελτιώσεων, κυρίως όσον αφορά τα δεδομένα που χρειάζονται να καταθέσουν οι πολίτες όταν υπογράφουν η πρωτοβουλία πολιτών ανάλογα με το κράτος μέλος, την χρονική διάρκεια της διαδικασίας για τη συλλογή των ή, ή το θέμα της συλλογής ε, διαγραμμικά, μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, των υπογραφών. Η Επιτροπή βεβαίως ε, είναι δεσμευμένη εξασφάλιση μιας επιτυχούς λειτουργίας πρωτοβουλίας των πολιτών. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχει ειμαστε επισημενοι δυναμικό ώστε να επανασυνδέσει τον πολιτή με τα θεσμικά τους όργανα. Επίσης, Θέλουμε να συζητήσουμε στου επόμενου μήνε και επί τη βάση τη εκθέσεώ μα με όλου του εμπλεκόμενου φορεί και τα λοιπά θεσμικά όργανα τον τρόπο βελτίωση αυτού του σημαντικού εργαλείου. Εν προκειμένου, εν προκειμένου καλωσορίζουμε την ε, ε, σύνταξη, όπως την επικείμενη σύνταξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια εκθεστία πρωτοβουλία ω απάντηση στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονό ότι ήδη έχει ξεκινήσει να συζητάει το θέμα αυτό και το Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που γύρονται με την έκθεσή μα είναι η ανάγκη να εξασφαλιστούν ότι θα ακούγονται οι διαφορετικέ θέσει και υπόψεις κατά τη διάρκεια μια δημόσια ακρόαση, Η τριμηνιαία περίοδο ε, που προβλέπεται ώστε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση σχέση με την πρωτοβουλία είναι πολύ σύντομη και η δημόσια αυτή ακρόαση επιτρέπει την συλλογή των διαφορετικών θέσεων πάνω στο θέμα αυτό. Επιπλέον λοιπόν και πέραν το ότι παραμένουν οι κύριοι πρωταγωνιστές στη διαδικασία αυτή, οι έχοντες την πρωτοβουλία, οι οργανωτές πρωτοβουλίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις και τριών εμπειρογνωμόνων στο θέμα αυτό σήμερα. Του έχει προσκαλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια καινοτομία που καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ε, τρέχουσα πρακτική και στο μέλλον για τις λοιπές πρωτοβουλίες πολιτών. Θα θέλω λοιπόν να καλωσορίσω και τους ε, ε, διοργανωτές της πρωτοβουλίας καθώς ε, και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και το Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών γιατί επιτρέπει να εξεταστεί ένα πολύ λεπτό και σημαντικό ζήτημα και δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα όλες τις προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προωθήσουν οι στόχοι όπως έχουν εγγραφεί στη συνθήκη. Έχουμε συναντηθεί με τους οργανωτές σε μια χωριστή συνεδρία που μας επέτρεψε να αντιληφθούμε καλύτερα τις ανησυχίες τους ε, με το συγκεκριμένο αίτημα που ήταν να καταργηθεί ή, ή μάλλον να ακυρωθεί η οδηγία 2010-63 για την προστασία των ζώων. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσεκτική την ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει και Βεβαίως θα ακούσετε και τον Γενικό Διευθυντή Καρλ Φάλκενμπεργκ από τη Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει πολύ σύντομα την κατάσταση σε σχέση με την οδηγία 2010-63 για τις δοκιμές της ζώα, το νομικό της Υπόδραφου του στόχου της και την κατάσταση σχέση με την υλοποίησή της. Βέβαια καταγράφουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές θέσει όπως θα εκφραστούν σήμερα το απόγευμα. Θα, ακολουθήσουμε, θα παρακολουθήσουμε μεγάλη προσοχή όλα τα διαφορετικά επιχειρήματα που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στο να διευκρινιστεί ακόμη περισσότερη κατάσταση. Κατόπιν της ακροάσεως και λαμβανομένων υπόψη των διαφορών θέσεων και επιχειρημάτων, η Επιτροπή θα ετοιμάσει την επίσημη απάντησή της στην πρωτοβουλία πολιτών στο Vivisection, ε, την οποία απόφαση προβλέπεται να υιοθετήσουμε στις 3 Ιουνίου, προκειμένου να τηρηθεί και η τριμηνία προθεσμία, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, λέει ο ομιλητής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα δίνω το λόγο στους οργανωτές. για να μας παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους. Ράις. Ταμίνο, Ο κύριος Στομένα και ο κύριος Ράις θα κάνουν την παρουσίαση. Θα μιλήσω την Ιταλική για να εκφραστώ ορθότερα χρησιμοποιώντας τη μητρική μου γλώσσα. Να ξεκινήσω από μία σκέψη που ακούγεται συχνά ότι το θέμα των πειραμάτων σε ζώα είναι ένα θέμα θα έλεγα δεοντολογικό, ένα θέμα ηθικό για την προστασία των ζώων. Βασικός μας στόχος ως οργανωτών αυτής της πρωτοβουλίας είναι το να προσπαθήσουμε να δούμε εάν η χρήση στα πειράματα αυτά των των ζώων είναι χρήσιμη για λόγους υγείας των πολιτών Δηλαδή βασικός μας στόχος είναι να αναρωτηθούμε αν σήμερα επιστημονικά η χρήση πειραμάτων σε ζώντα ζώα δίδει εγγυήσει στους Ευρωπαίους πολίτες στον τομέα της υγείας. Και η απάντησή μας είναι όχι, αλλά δεν είναι η δική μας απάντηση αυτή. Είναι η απάντηση πολλών α, ε, μεταναλυτών επιστημόνων οι οποίοι απέδειξαν ότι ένα τεράστιο ποσό αξιολογήσεων στις έρευνες που έχουν γίνει με πειράματα στα ζώα αποδεικνύουν ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις στα πλαίσια των οποίων δεν υπάρχει αναλογία ανάμεσα σε αυτά τα οποία βρίσκει κανείς όταν κάνει πειράματα στον άνθρωπο και όταν κάνει πειράματα στο ζώο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα ζώο σαν πρότυπο για πειράματα σε άλλα ζώα. Όταν εμείς αναφερόμαστε στα τροπτικά <coughs> βλέπουμε ότι η αντιστοιχεία των αποτελεσμάτων και των στοιχείων ανάμεσα στον ποντικό από τη μία και τον αρουραίο από την άλλη δεν ξεπερνά το 50%. Πώς μπορεί κανείς να, ε, να βασιστεί σε τέτοιες συγκρίσεις με το ανθρώπινο όν όταν υπάρχει μια διαφορά 50% απέναντι σε, ανάμεσα σε δύο τόσο κοντινά ζώα. Λοιπόν, τι είναι σωστό σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς ξέρω ότι για να εγκρίνω μια διαδικασία ιατρική πρέπει να την ελέγξω στον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση ε, μέσω των πειραμάτων σε άλλα είδη, σε άλλα ζώα και σε επίπεδο τεξουσικολογικό. Σκεφτείτε λίγο τον κανονισμό REACH που σε επίπεδο χρήσης των ζώων δεν δίδει και δεν δέχεται εγγυήσει από πειράματα με ουσίες που περιλαμβάνονται στο ρίτς στα ζώα. Αν πραγματικά θέλαμε να έχουμε ε, διάφορες ε, στρεβλώσεις στις γεννήσεις των ζώων και προβλήματα ιατρικά, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά στοιχεία που μας επιτρέπουν να ε, δούμε ε, ποιες είναι οι τοξικές ουσίες, οι καρκινογόνες ουσίες. Έχουμε φτάσει γύρω στις 20.000 θεωρητικά. Δεν μπορούμε να βρούμε μεθόδους για όλες αυτές συνολικά, αλλά ούτε και για κάθε μία ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε τρόπους οι οποίοι να είναι έγκυροι και έγκριτοι και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του περιβάλλοντος, τον σεβασμό των κανονισμών, την προστασία των ζώων και κυρίως την προστασία των ανθρώπων. Συνεπώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει συλλέξει αυτόν τον ιδιαίτερα υψηλό υπογραφών από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών Έχουμε ένα εκατομμύριο χιλιάδες υπογραφές αν λάβουμε υπόψη μας και αυτές οι οποίες για διάφορους τρόπους λόγους δεν ελήφθησαν υπόψη. Και αν προσπαθούμε να δούμε σήμερα την κατάσταση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών ξέρουμε ότι δεν υπάρχει και σε καμία περίπτωση αντιστοιχεία ανάμεσα στο είδος της έρευνας η οποία γίνεται και στο επίπεδο προστασίας. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι όγκοι στα παιδιά σαν παράδειγμα ή αυξάνονται οι ψυχολογικές ασθένειες στους ηλικιωμένους, οι εκφυλιστικές ασθένειες στους ηλικιωμένους. Και τα πειράματα στα ζώα δεν έχουν δώσει σε καμία περίπτωση ικανοποιητικές απαντήσεις. Αυτό το οποίο ζητάμε λοιπόν είναι να υπάρξει μια κάποια διαφάνεια αν το σύστημα αυτό ε, των ε, ε, πειραμάτων στα ζώα είναι προληπτικό με την έννοια της πρόβλεψης περισσότερο για αντίστοιχες καταστάσεις στον άνθρωπο. Όχι. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα μεθόδους περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, επενδύοντας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και δίδοντας πραγματικές εγγυήσεις, κατάλληλες εγγυήσεις στα εργαστήρια να χρησιμοποιούν μεθόδους πιστοποιημένες, έγκυρες, σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις προβλέψεις της συνθήκες μας. Εάν προβλέπει η συνθήκη την εγγύηση της υγείας των πολιτών, η μέθοδος αυτή με πειράματα στα ζώα δεν το κάνει Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να γίνουν περισσότερες έρευνες εκτός αυτών. Η μεγάλη ποσότητα των εργαστηριακών μεθόδων που υπάρχουν στην λογοτεχνία σε εισαγωγικά την επιστημονική έχουν επικυρωθεί και έχουν μάλιστα επικυρωθεί επιστημονικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρουμε σε έναν κατάλογο που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκατοντάδες περιπτώσεων επιστημονικής βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν τις δικές μας θέσεις και για τη μη εγκυρότητα των πειραμάτων σε ζώα και για τη μη προβλεψιμότητα και για την δυνατότητα χρήσης μεθόδων αντικατάστασης. Και όταν μιλάμε για αντικατάσταση δεν μιλάμε για μεθόδους με λιγότερα ζώα αλλά μιλάμε για μεθόδους χωρίς ζώα. Είναι σαφές ότι σε μια τέτοια ακρόαση δεν έχουμε το χρόνο για να κάνουμε μια πλήρη επιστημονική παρουσίαση μέσα σε ένα επτάλεπτο. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, να τα θέσουμε στην διάθεση του Κοινοβουλίου και στην διάθεση της Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αν πράγματι υπάρχει μία μέθοδος πιο έγκυρη από αυτήν που μας παρουσιάζουν σήμερα για να εγγυηθούμε την υγεία των πολιτών με επιστημονικό τρόπο και στον τοξικολογικό τομέα και στον τομέα τον φαρμακολογικό. Και γενικά βλέπουμε ε, στους τομείς ε, στους οποίους οι ρυθμίσεις οι κοινοτικές προβλέπουν και τη χρήση των ζώων όπως τα ε, εντομοκτώνα, στα, τροφι, στα πρόσθετα, στα τρόφιμα κτλ αυτό το κομμάτι θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να δοθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στον Ευρωπαίο πολίτη. Panie Rajs, czas dla Pana. 7 minuty. Oui, euh, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε για να πάρουμε μέρος σε αυτήν την αντιπαράθεση ιδεών. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μέχρι τώρα οι κανονισμοί που αφορούσαν τα πειράματα μετά από την ε, διάσκεψη της Λισαβόνας ήταν δεδομένα. Είχα παρουσιάσει στα αγγλικά την προεστήμασία μου και θα σας ε, μιλήσω τελικά ε, χωρίς έγγραφο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσκλησή της. Λέγομαι Κλόντρες, ήμουν διευθυντής στο ΣΕΝΕΡΕΣ για τέσσερα χρόνια και δραστηριοποιούμε στον τομέα της βιολογίας εδώ και 60 χρόνια. Οι μη, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ε, έχουν συνυπογράψει αυτή την ε, συλλογή ε, υπογραφών ε, θυμίζω ότι έχουν υπογράψει πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι την πρόταση αυτή, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα εκατομμύρια που συμμετέχουν στις εργασίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων που πήραν την πρωτοβουλία. Εμείς θέλουμε να αμφισβητήσουμε την 63 του 2010 που λέει ότι τα ζώα είναι προβλέψιμη βάση, πλατφόρμα για πειράματα σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών είναι αποδεκτά. Ε, φυσικά δεν συμφωνούμε με αυτό εμείς. Ένα ζώο ε, ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα βιολογικό πρότυπο για κάποιο άλλο. Κανένα είδος δεν είναι πρότυπο για κάποιο άλλο. Θα μου πείτε αυτή είναι μια θεωρητική παρατήρηση. Όχι, θα σας το αποδείξω μαθηματικά. Τι καθορίζει ένα είδος καταρχάς ένα είδος ε, είναι θωρακισμένο θα έλεγα. Αυτό σημαίνει καταρχάς απομονωμένη ε, αναπαραγωγική διαδικασία. Γάτα με σκύλο δεν πηγαίνει. Ε, επίσης η κληρονομιά, η γενετική είναι μοναδική και ενιαία. Αμφισβητείται όταν υφίσταται κάποιο στρες το συγκεκριμένο είδος, μια συγκεκριμένη αμφισβήτηση όπως σε έκθεση σε ασθένειες, σε χημικά προϊόντα, χιλιάδες εν πάση επιθέσεις και που δημιουργούν προβλήματα στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, κάθε είδος θα αντιδράσει με το δικό του ADN, με τα δικά του γονίδια, και ένα άλλο είδος το οποίο έχει μια διαφορετική γενετική κληρονομιά θα χρησιμοποιήσει διαφορετικά γονίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξουν ε, όμοιες αντιδράσεις. Μπορεί να μοιάζουν ή μπορεί να είναι αντίθετες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα είδος είναι πρότυπο για τα υπόλοιπα βιολογικά αξιόπιστο. Και αυτό ισχύει και για την πρόληψη στον τομέα της υγείας γενικότερα και για την υγεία την ανθρώπινη και για την ιατρική έρευνα. Αυτό παρουσιάζει βέβαια μια μεγάλη ευκολία για τη χημική βιομηχανία. Αν έχετε ένα προϊόν χιν και θέλετε να το βάλετε στην αγορά και είναι ο λίγων καρκινογόνο το προϊόν σας. Για να αποδείξετε ότι δεν είναι καρκινογόνο ή ελάχιστα επιλέγετε μια γραμμή ε, ποντικών σαν παράδειγμα την 67-1, η οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτική σε σχέση με επιθέσεις καρκινογόνων. Αν χρησιμοποιήσετε όμως μία άλλη γραμμή καταγωγής η οποία είναι πολύ ευάλωτη στην ανάπτυξη καρκίνων του στήθους τότε προφανώς τα πειράματα με το ίδιο προϊόν δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Το ίδιο και με τα ιστρογόνα. Ε, αν το χρησιμοποιήσετε στα C1H H, ειναι εντελώς διαφορετικά τα αποτελέσματα από το, 50, ε, από το 50, Β53 κάθετος 6. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ναι μεν έχει μια ευκολία ο βιομήχανος αλλά οι συνέπειες είναι σοβερές καταστροφικές στον τομέα της υγείας και σε σχέση με τις επιπτώσεις και σε σχέση με την επιβολή ασθενειών όπως ο διαβήτης, το αλτσχάιμερ, ο καρκίνος και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καρκίνος του στήθους ή ο καρκίνος του προστάτη όπως επίσης και ο αυτισμός. Δυστυχώς θα ήθελα να σας δείξω κάποιους, κάποια γραφήματα με αριθμούς στοιχείων που συλλέξαμε στη Γαλλία με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας αλλά δεν μπόρεσα να κατεβάσω από το ίντερνετ γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε βάσεις δεδομένων εξωτερικές από μέσα από το κοινοβούλιο. Από το 9 λοιπόν και μετά και με βάση τα στοιχεία γαλλικών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα δημόσιας υγείας, ο διαβήτης, τα συμπτώματα έχουν ε, διπλασιαστεί σε 9 χρόνια. Το Alzheimer σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Ε, ο καρκίνος του στήθους πάνω ε, από 50%, ο, προστάτης, ο καρκίνος του προστάτη κατά 50%, και ο αυτισμός κατά 50% από το 2000 μέχρι το 2009 και ο αριθμός αυτών που ζουν με την ασθένεια έχει αυξηθεί 250 ή 300 φορές. Εκτιθέμεθα δηλαδή συστηματικά σε προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά. Αν συνεχίσουμε με τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα τότε τα παιδιά μας που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά όταν γίνουν ενήλικοι το 2050 ο ένας στους τρεις θα είναι διαβητικός, ο ένας στους τέσσερις θα υποφέρει από Αλσχάιμερ, μία γυναίκα στις τρεις θα υποφέρει από καρκίνο στο στήθος, ένα μεγάλο ποσοστό ε, των ανδρών θα υποφέρει από καρκίνο του προστάτη και ε, ε, θα υπάρχει μία γέννηση με αυτιστικό παιδί στις τρεις γεννήσεις και μιλάμε τώρα για σε 50 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τον πειραματισμό μέσω των ζώων, τα πειράματα μέσα από τα ζώα. Έχει υπάρξει σημαντική επιστημονική πρόοδος τα τελευταία 20-30 χρόνια και οι μέθοδοι αυτοί μας δίνουν κάποιες, ε, κάποιες, ε, κάποια στοιχεία για την αξιολόγηση της τοξικότητας των προϊόντων. Έχουμε σαν παράδειγμα σε σχέση με τα ε, ισχυρά κύτταρα, τα IPS, τα πολυδύναμα ίσως κύτταρα, αρκετά νέα στοιχεία. Μπορούμε να παίρνουμε τα κύτταρα αυτά χωρίς να δημιουργούμε βλάβη στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή είδος από τα έμβρια, από τα παιδιά, από τα νέα παιδιά, από τους ενήλικες, από τους ε, ηλικιωμένους και μπορούμε να διαφοροποιούμε και ανάλογα με την ε, φυλή στην οποία ανήκουν τα πρόσωπα αυτά και οι μέθοδοι αυτοί επιτρόπουν λοιπόν να εξετάζουμε ε, τα κύτταρα αυτά με ένα χημικό προϊόν σε μια χρονική διάρκεια και με μια πυκνότητα προαπαιτούμενη έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα που εφαρμόζονται συνολικά σε μας. Ένα κύτταρο φυσικά δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μπορούμε εμείς τις μελέτες αυτές να τις μεταφέρουμε από τα κύτταρα σε ιστούς μέσω... Α μέσω χορήγησης υδρών, εν περιπτώσει στο αίμα. Και μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε ε, σε ε, παραγωγή αποτελεσμάτων όπως το απαιτεί το ΡΙΤΣ που θεωρεί ότι το ΡΙΤΣ βέβαια ότι πρέπει να γίνουν τα πειράματα στα ποντίκια. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Αυτά λοιπόν για την αξιολόγηση των τοξικολογικών κινδύνων για την βιοιατρική έρευνα. Θα αναφερθώ σε ένα βραβείο Νόμπελ, το Σίδνεϊ Μπράιερ, που λέει ότι θα πρέπει να γίνεται η έρευνα στην βιολογία από την κούνια μια τελευταία φράση. Δεν είναι παραδοσιακή ακρόαση γιατί έχουμε πολλά όρια χρονικά περιορισμούς χρονικούς. Πάντως δεν πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει, πρέπει να αλλάξουμε ρυθμό. Η βιολογική έρευνα γενικά έχει σημειώσει σημαντικότατες προόδους. Έχουμε πάρα πολλές τεχνικές, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, που μας επιτρέπουν να δώσουμε απαντήσεις ε, ε, στην ανθρώπινη υγεία ανεξαρτήτως των ζώων i przepraszam za swoją bardzo... ευχαριστώ πολύ. Στο συγγνώμη αν σας διακόπτω, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας Προέδρου. Να πω ότι μεταδίδεται και ζωντανά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας αυτή η ακρόαση και τώρα να περάσουμε σε μια άλλη παρουσίαση συγκεκριμένα από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος λοιπόν Φάλκενμπεργκ, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, να καθίσετε στο βήμα. Χαιρετίζουμε τον κύριο Κατάν, τον Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Η Ευρώπη έχει ένα από τα πιο προηγμένα νομικά πλαίσια για την προστασία των ζώντων ζώων και γι' αυτό είναι και ένα πλαίσιο το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε την οδηγία για την προστασία των ζώντων ζώων. Επτά χρόνια πήρε μέχρι να καταρτιστεί. Έχουμε τώρα ένα συμβιβασμό. Δεν είναι κανοπιτικός για κανέναν, αλλά όπως ήθεστε να λέγεται, ένα συμβασμό είναι καλό όταν δεν είναι κανείς ικανοποιημένος με αυτόν. Τώρα, τα ζητήματα τα οποία έχουν ε, θέσει οι συμπολίτε μα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και να τα λάβουμε υπόψη μα. Ε, Αυτό κάνουμε και τώρα. Εξετάζουμε, θα καταλήξουμε σε κάποια απορίσματα, Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φάλκεμπεργκ για να μας δώσει το υπόβαθρο και το ιστορικό του ρυθμιστικού αυτού Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που διοργανώσατε την ακρόαση αυτή. Θέλω να πω ότι νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκω μεταξύ τόσων γνωστών εξεχόντων ε, επιστημόνων. Εγώ που οικονομικά έχω σπουδάσει μόνο, αλλά αφού με καλέσατε για να σας κάνω μια παρουσίαση του ρυθμιστικού πλαισίου της ρυθμιστικής πραγματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να το κάνω γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και γι' αυτό θα εστιάσω ενδεχομένω σε κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένα από αυτά τα θέματα που ακούσαμε μέχρι τώρα. Έχουμε τη βασική πρόταση της ε, πρωτοβουλίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απόκληση απόψεων ως προς αυτή τη βασική θέση. Όλοι είμαστε πεπισμένοι, πιστεύω, ότι πολύ καλύτερες και ασφαλέστερες μέθοδοι και δοκιμές μπορούν να αναπτυχθούν. Ορισμένες εξ αυτών ήδη οριμάζουν το ε, στην αγορά σε σχέση με παραδοσιακές δοκιμές και πειράματα σε ζώα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέτασε την νομοθεσία της σχετική το 86 συγκεκριμένα και καταλήξαμε στην οδηγία 63 του 2010. Με την οδηγία αυτή ουσιαστικά δεν επιβάλλεται η μέθοδος ε, της χρήσης ζώντων ζώων για πειράματα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να, είναι, ε, να χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 λέγεται ότι τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι όποτε είναι δυνατόν χρησιμοποιείται αντί της διαδικασίας άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμή χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου. Χρησιμοποιείται. Το επαναλαμβάνω αυτό αντί της διαδικασίας. Διαδικασία στη γλώσσα μας, την επιστημονική αυτή αργό ας πούμε, είναι ουσιαστικά το πείραμα ή δοκιμή πάνω σε ένα ε, ζώο. Άρα λέει ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν άλλες επιστημονικά ικανοποιητικές μεθόδους ή δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων. Και θα πρέπει να διασφαλίσετε από τα κράτη-μέλη ότι θα γίνεται αυτό η νομοθεσία αυτή. Το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στο βήμα προηγουμένως έχει μεταφερθεί επιτυχημένα στο εθνικό δίκαιο και των 27 κρατών μελών, όμως είναι σχετικά πρόσφατο νομοθέτημα. Δηλαδή άρχισε να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη από τα τέλη του 2013. Επομένως, η εμπειρία και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού είναι πρόσφατα σχετικά και θα αντλήσουμε ουσιαστικά τα πρώτα διδάγματα στην πρώτη έκθεση που θα καταρτήσουμε πέντε χρόνια μετά την έναξη εφαρμογή στο 2018 κάθετος 19 θα παρουσιάσουμε το σχετικό κείμενο πλήρη δηλαδή αναθεώρηση της εφαρμογής οδηγίας θα την υποβάλουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η οδηγία πέραν αυτού του άρθρου που σας ανέφερα, που ουσιαστικά απαιτεί την ε, χρήση εναλλακτικών μεθόδων όταν αυτές δεν έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί, έχει ως στόχο ότι η χρήση των ζώων σε παραδοσιακές διαδικασίες ε, μειώνεται, πρέπει να μειωθεί. Αν δούμε τις προϋποθέσεις και τους όρους Βλέπετε ότι αυτό που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε είναι στα εργαστήρια τα ζώα τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές να την χάνουν τις πλέον αξιοπρεπούς δυνατής μεταχείρισης να μειωθεί δηλαδή ο πόνος, τα λεπορία, η αγωνία τους κτλ. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίζουν τα κρατη Θεωρούμε λοιπόν ότι η πραγματική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να επικυρώσουμε γρήγορα άλλες ε, μεθόδους δοκιμών, ώστε στον πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία του 2010 να μπορούμε αυτές τις νέες ε, μεθόδους να μεθόδου, να τις επιβάλλουμε του εικόνε, να τις καταστήσουμε υποχρεωτικές ε, στα εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα προηγείται σε μεγάλο βαθμό οποιοδήποτε άλλο κράτους ε, στον πλανήτη που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ε, εταίρος, σε σημαντικούς μας εταίρους, που να έχει στην νομοθεσία του τόσο ξεκάθαρη ρήτρες υπέρ της προστασίας της ευζοίας των ζώων. Ούτε που να απαιτεί ρητός τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων όποτε αυτό είναι δυνατό. Στην πραγματική ζωή και νομίζω ότι μεγάλο μέρος ε, της κριτικής που ακούσαμε εδώ, από εκεί προέρχεται, στην πραγματική ζωή οι επιστημονικές επιτροπές έχουν καταλήξει, άκουσα τις παρουσιάσεις και είμαι βέβαιος ότι έγιναν καλή την πίστη όταν βλέπουμε τις επιστημονικές επιτροπές να συζητούν αυτά τα θέματα, ξεκολουθούμε δυστυχώς να ακούμε να τίθεται υπό αμφισβήτηση εγκυρότητα κάποιων επιχειρημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνει στις συνθήκες ε, την ευζοία και την καλή μεταχείριση των ζώων ως στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και αρχή της προφύλαξης που και αυτή κατοχυρώνει τις συνθήκες. Και νομίζω ότι συλλογικά αυτό που πρέπει να δουλέψουμε και ελπίζω να συνεισφέρει ως προς αυτό το στόχο και η Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία είναι πιο αποφασιστικά και πιο γρήγορα να καταλήξουμε σε επιστημονικές συμφωνίες ως προς τις διαδικασίες οι οποίες είναι επαρκώς έγκυρες, σταθερές, θέρες για να μπορούμε να τις εμπιστευτούμε. Άκουσα ε, επαναλημμένως στην ακρόαση ότι το REACH απαιτεί τις δοκιμές σε ζώο. Ναι, αυτό αληθεύει, αλλά ως τελευταία λύση. Το REACH, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος δοκιμών, απαιτεί τη χρήση εναλλακτικών μέτρων υφιστάμενα δεδομένα και μόνο σε έσχατη λύση και αν δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα αποδέχεται και τα πειράματα σε ζώα, τις δοκιμές σε ζώα. Αυτό το λένε οι κανονισμοί. Λογικά, λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να γίνει και πραγματικότητα στα εργαστήρια των χωρών μας. Αλλά και στους επιστημονικούς φορείς που έχουμε συγκροτήσει για να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες αυτές τις οποίες έρχονται σε επαφή οι πολίτες μας καθημερινά με το σωστό τρόπο και με τη λιγότερη προσφυγή σε πειράματα σε ζώα έχουν ελεγχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, θα χαρούμε πολύ αν μπορέσετε να παραμείνετε για να παρακολουθήσετε την ακρόασή μας. Τώρα καλό τον πρώτο ειδικό, τον κύριο Γκουίκ. Να λάβει το λόγο. Πριν όμως ξεκινήσετε, θα ήθελα να πω ότι αφού γίνει η πρώτη παρουσίαση, θα γίνει μια, ε, ένας γύρος αποκρίσεων από τους βουλευτές, όσους ε, ζήτησαν να λάβουν το λόγο. Στη συνέχεια, με διαδικασία κάτι όποιος δηλαδή προλάβει να στήσει το λόγο, εάν υπάρξει χρόνος. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρεμενάς και Εάν ο προσκεκλημένος μας, κύριος Ray Greek, είναι έτοιμος, με πολύ μεγάλη χαρά θα του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Is the uh, microphone functional? Yeah. Good. Excellent. Thank you. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας που μου επέτρεψαν να πάρω το λόγο σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλες τις ΜΚΟ που με έφεραν εδώ. Είναι πάρα πολλές, δεν μπορώ να τις αναφέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε παρόντες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το να μπορέσω να πάρω το λόγο μπροστά σας προσεκλήθην λόγω της εμπειρίας μου που έχω στην προτυποποίηση των ειδών. Έχω πάνω από 20 δημοσιεύσεις που ασκούν κριτική στα πρότυπα τα οποία αποκολουθούμε μέχρι σήμερα. Αυτά δεν είναι άρθρα που αφορούν με αποτελέσματα ερευνών, αλλά άρθρα που αμφισβητούν την φιλοσοφία της επιστήμης η οποία στηρίζει αυτού του είδους τις αντιλήψεις. Είμαι εμπειρογνώμων στην προτυποποίηση των ζώων και όχι στην χρήση ενός ζώου για συγκεκριμένη ασθένεια κάθε φορά. Έχω συγγράψει αρκετά βιβλία, κεφάλαια, άρθρα, επιστημονικά, μέσα ενημέρωσης. Έχω δώσει ομιλίες στον κόσμο υπέρ το, μάλλον για τα υπέρ και τα κατά. Υπάρχουν και υπέρ. Ήμουν καθηγητής σε δύο πανεπιστήμια στις Ηνωμένε Πολιτείες και δεν έχω οικονομικά ωφέλη από την κατάληξη αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν θα με επηρεάσει οικονομικά ή αλλώς. Ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρομαι είναι γιατί πάρα πολλοί αναφέρονται σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και λένε ότι όλοι οι επιστήμονες υποστηρίζουν τη χρήση των ζώων. Οι έρευνες αυτές είναι παραπλανητικές γιατί όλοι συνήθως έχουν οικονομικά συμφέροντα και δεύτερον οι μελέτες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα στο οποίο εγώ ε, παρεμβαίνω, δηλαδή την προβλεπτική δυνατότητα που έχουν κάποιες συγκεκριμένες μέθοδες. Η επιστημονική κοινότητα και η φαρμακευτική κοινότητα υποστηρίζουν ότι τα πειράματα έχουν άμεση σχέση με την υγεία των ε, ε, ανθρώπων και των ζώων. Υπάρχουν 180 εμβόλια για το AIDS, τα οποία απέδωσαν σε σχέση με τα ζώα, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν επιτυχές ε, για τους ανθρώπους. Ούτε ένα στα εκατό. Οπότε πώς μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων. Είδαμε χίλια περίπου φάρμακα νευροβιολογικά και εκεί ε, είχαν αποδώσει στα ζώα αλλά κανένα δεν μπόρεσε να περάσει στην αγορά των, ε, ε, των ανθρωποφαρμάκων. Λοιπόν, υπάρχει μια πλήρης έλλειψη, αν θέλετε, χρησιμότητας της χρήσης ζώων για την προστασία του ανθρώπου. Αυτό είναι ο με τον οποίο εγώ ασχολούμαι. Η προβλεπτική αξία, αν θέλετε, είναι η βασική ε, αιτία χρήσης των ζώων. Και είναι κάτι το οποίο... Χρησιμοποιούνται εδώ και με εννέα, τρόπου, ε, τρόπους ε, τα ζώα στην επιστήμη. Καταρχάς χρησιμοποιούνται σαν προβλεπτικά πρότυπα για ασθένειες, για τον έλεγχο των φαρμακευτικών ουσιών. Ε, φυσικά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ένα ζώο σαν πηγή απλά η ινσουλίνης ή να μάθει πράγματα για τη φύση. Από το 3 μέχρι το 9 υπάρχουν μένα, αλλά υπάρχουν και πολλές εναλλακτικέ σήμερα. Δεν ίσχυε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό πρόβλημα είναι με το 1 και το 2. Το 1 και το 2 δείχνουν το πώς η έρευνα σε ζώα πωλείται στην κοινωνία, περνάει στην κοινωνία. Υπάρχουν δύο βασικές αρχές της επιστήμης που ακυρώνουν την χρησιμότητα των ζώων. Το πρώτο είναι η εξέλιξη. Πρόκειται εδώ για έναν πίνακα ο οποίος δείχνει πως ε, οι πρόγονείς μας ε, οδήγησαν ε, στους ουραγκοτάγκους, στους γίβονες, τις μαϊμούδες, τους γορίλες, τους χιμπατζίδες κτλ. Έχουμε κάποια κοινά γενετικά στοιχεία, αλλά με το χρόνο έχουμε αποκλίνει από την κοινότητα αυτή. Οι διαφορές αυτές δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι αρκετά μικρές. Ο δεύτερος τομέας της επιστήμης που ακυρώνει την χρησιμότητα των ζώων είναι η γνωστή επιστήμη ως επιστήμη της περιπλοκότητας. Βλέπετε αυτήν την διαφάνεια πάρα πολύ περίπλοκη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Έχω βάλει όμως τρεις κύκλους τους οποίους θα ήθελα να σταθείτε ένα περίπλοκο σύστημα αποτελείται από απλά συστήματα τα οποία υπάρχουν σε χαμηλότερα επίπεδα οργάνωσης. Δηλαδή ξεκινάμε από την σκόνη, ε, οξυγόνο, υδρογόνο, άνθρακας και αυτό είναι ένα περιβάλλον που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στον άνθρωπο, στα κοτόπουλα ή σε άλλα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία συνδυασμένα δημιουργούν γονίδια και τα γονίδια συνδυασμένα δημιουργούν συστήματα και φτάνουμε σε υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης όπου εκεί πια τα περίπλοκα αυτά συστήματα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Και επειδή ακριβώς λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, δημιουργούν χαοτικές συνθήκες. Και εδώ έρχεται η θεωρία του χάους. Έχετε εδώ ένα μαθηματικό πρότυπο. Βλέπετε ότι ένα περίπλοκο σύστημα διαφέρει από ένα δεύτερο περίπλοκο σύστημα μόνο κατά την τέταρτη θέση και πέρα. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή διαφορά από ένα σημείο και μετά μόνον. Όπως βλέπετε εδώ οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην ανοιχτόχρωμη γραμμή και στην σκουρόχρωμη γραμμή γίνεται ολοένα και περισσότερο εμφανής. Αυτό σημαίνει ότι αν δώσετε ένα φάρμακο σε ένα άνθρωπο την μαύρη γραμμή τότε θα σκοτώσει τον άνθρωπο. Αν δώσετε όμως στον άνθρωπο την γκρίζα γραμμή τότε το φάρμακο θα λειτουργήσει θεραπευτικά. Αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι συμβαίνει στην ανθρώπινη ιατρική. Δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο τρόπο στις ασθένειες και στα φάρμακα. Τέλος, για να στηρίξει κανείς τις θεωρητικές μας ανησυχίες, μιας και προέρχομαι από τη θεωρία και την επιστήμη της περιπλοκότητας, υπάρχουν και εμπειρικές παρατηρήσεις για τη μη χρησιμότητα των τεστ σε ζώα. Εδώ βλέπετε μία διαφάνεια, υπάρχουν πάρα πολλές στην ε, επιστημονική τεκμηρίωση για πολλά θέματα, αλλά η συγκεκριμένη αυτή η διαφάνεια διαπιστώνει την βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων σε τρία είδη ζώων, στους πυφίκους, στα ερπετά και στα σκυλιά και στον άνθρωπο από την άλλη βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα στην οργάνωση του γραφήματος. Εμείς αυτό το λέμε ε, μια πολυδιασπασμένη, αν θέλετε, σαν τα σκάγια της βολής γραφή, ε, παρουσίαση μέσω γραφήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα ε, διάφορα όργανα επηρεάζονται με, διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους. Εάν υπήρχε δυνατότητα χρήσης προβλεπτικής των ζώων, τότε θα έπρεπε να υπάρχει μία ομοιότητα και θα έπρεπε να υπάρχει μία γραμμή, μία γωνία 45 μοιρών από το κάτω μέρος προς τα πάνω, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτό το ε, γράφημα. Ακόμα και αν κάποια ζώα έχουν μία αντίστοιχη εν μέρη τουλάχιστον βιοδιαθεσιμότητα, ε, τα δεδομένα αυτά δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε σε βάθος ε, το, τη σχέση τους ε, με τον άνθρωπο. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τοξικά, τοξικές ουσίες και για καρκινογόνες ουσίες κτλ. Και γι' αυτό ακριβώ τον λόγο δυστυχώς όμως χρησιμοποιούμε τα ζώα για να ερευνούμε το τι θα γίνει στον άνθρωπο άμα του δοθεί μια κάποια ουσία. Έχουμε αποτύχει πλήρως εδώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούμε τις μεθόδους αυτές, δυστυχώς. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι και τα ζώα δεν έχουν τίποτα κοινό. Έχουν κοινά στοιχεία. Όλα τα θηλαστικά έχουν πνεύμονες, έχουν καρδιές και τα όργανα αυτά κάνουν την ίδια περίπου δουλειά αλλά οι ασθένειες προκαλούν εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις από αυτές τις υψηλά περίπλοκες μορφές οργάνωσης, σωματικής οργάνωσης. Και οι ανομοιότητες ε, ε, υπερισχύουν των ομοιοτήτων όχι μόνο υπάρχουν ε, διαφορές γενετικές, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλου τύπου διαφορές οι οποίες οδηγούν σε τεράστιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Σήμερα ζούμε τη λεγόμενη προσωποποιημένη ιατρική. Θέλουμε δηλαδή να ταιριάξει το φάρμακο ε, με τα γονίδια του ασθενούς, όχι με τα γονίδια της μαμάς του ή του παππού του. Δεν υπάρχει ένα νούμερο που να κάνει για όλους μια συνταγή καλή για όλους. Ξέρουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες αντιδρούν διαφορετικά στις ασθένειες και ε, στα φάρμακα όπως και οι εθνοτικές ομάδες επίσης. Είδαμε ότι ακόμα και οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι και αυτοί ακόμα διαφοροποιούνται στις ανταποκρίσεις, στις απαντήσεις τους στα φάρμακα και τις ασθένειες. Αν κάποιος σας πει ότι ένα πρότυπο ε, ζωικό έχει τροποποιηθεί γενετικά για να προσωμιώσει τον άνθρωπο, ρωτήστε τους ε, πόσο κοντά μπορεί να έρθει στον άνθρωπο όσο κοντά είναι δύο μονοζυγωτικοί δίδυμοι. Όταν δεν αντιδρούν οι δύο μονοζυγωτικοί με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο φάρμακο, τότε πόσο μπορεί να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο τα ζώα με τους ανθρώπους. Έχουμε επίσης εδώ και χρόνια την γνώση ότι πάρα πολλά φάρμακα δεν γίνονται ανεκτά από τους ανθρώπους. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Εσείς μου είπατε ότι έχω 16 λεπτά λέει ο μιλητές. Ζητώ συγγνώμη λέει ο κύριος Γκρίκ. Θα αφήσω κάποιες διαφάνειες γιατί δεν έχω πια πολύ χρόνο. Η πρωτοβουλία την οποία ασχολούμεθα σήμερα αφορά και την επιστήμη και τη δεοντολογία. Εάν πράγματι τα ζώα δεν έχουν δυνατότητα χρήσης τότε δεν πρέπει να θεωρείται ε, η μέθοδος των πειραμάτων σε ζώντα ζώα σαν αναγκαίο κακό. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Przechodzimy ευχαριστώ θερμά. Και τώρα περνάμε στην, ε, στο γύρο των ερωταποκρίσεων από τους συναδέλφους των ε, επιτροπών μας με χρόνο συγκεκριμένο σε όσους έχουν ήδη ζητήσει το λόγο. Έχουμε την κυρία Αγγιλέρα πρώτα. Δύο λεπτά το μέγιστον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ πολύ γρήγορα αυτούς που προωθούν αλλά και έχουν υπογράψει μέχρι τώρα την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκών Πολιτών που είναι πάρα πολύ θετική. Παρακολουθούμε την εξέλιξη με τη συλλογή υπογραφών και παρακολουθούμε και πολύ προσεκτικά και τις μέχρι τώρα παρουσιάσεις. Θα ήθελα επίσης εδώ να ευχαριστήσω όλους τους επιστήμονες, ερευνητές, όλους τους, διότι νομίζω ότι και όλοι όσοι έλαβαν το λόγο έχουν συνεισφέρει, αλλά και όλοι οι επιστήμονες και οι ερευνητές, ακόμη και όσοι πειραματίζονται μέσω, ε, βοηθούν ε, και βελτιώνουν την υγεία μας, βελτιώνουν την ποιότητα. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων, ε, δεν είμαι ειδική για την έρευνα ούτε για τα πειράματα σε ζώα. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να συλλέξω όλες τις δυνατές πληροφορίες. Ήρθα σε επαφή με ερευνητές, με επιστήμονες, ε, επισκέφθηκα και ένα κέντρο. Συγκεκριμένα το Τεχνολογικό Πάρκο Βιοιατρικής ε, στην Ισπανία, στη Γράδα και προσπαθώ όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες να συλλέξω. Όμως, έχω πραγματικά μεγάλες αμφιβολίες. Την οδηγία 63 του 2010, που λέτε ότι λέει ότι θα καταργηθούν αυτές οι διαδικασίες, ουσιαστικά ο στόχος της οδηγία αυτής ποιος είναι. Δηλαδή πλήρη αντικατάσταση των πειραμάτων σε ζώα. Κατά την άποψή μου είναι καλή αυτή η οδηγία κάτι λέτε, από βολική πλευρά δεν ε, μπορεί να υποκαταστήσει ένα ζώο ενό είδου σε ένα ζώο άλλου είδου. Έχω ακούσει και άλλα ε, αντίθετα επιχειρήματα. Δηλαδή, έχω ακούσει και τα δικά σα επιχειρήματα, αλλά και τα ακριβώ αντίθετα. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ψυχική αμφιβολία. Κατά τη δική μου άποψη σήμερα πολύ δύσκολα μπορεί να επικατασταθεί το πείραμα σε, στα ζωή, δοκιμές στα ζώα, εντελώς από άλλες μεθόδους. Νομίζω ότι είναι σωστή η εστίαση της οδηγίας. Ε, σίγουρα λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθούν τα πειράματα, αλλά δεν ξέρω εσείς όταν θα πάρετε το λόγο θα μπορούσατε να μου πείτε είναι πράγματι δυνατό να, να αντικατασταθούν απόλυτα όλα τα πειράματα, όλες οι δοκιμές σε ζώα. Κατά την άποψή δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βοητσεχόσκι, 1,5 λεπτό. Była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling. Ach, δεν φαίνεται να είναι εδώ. Χόισλινγκ, παρακαλώ, κύριο Χόισλινγκ. Ναι, πρόεδρο. Τι, δηλαδή τώρα έχω τρία Ε, ευχαριστώ πολύ έχοντας την πρωτοβουλία αυτής της πρωτοβουλίας. Βεβαίω ενημερωνόμαστε σήμερα με την ακρόαση και θα πρέπει μετά να γίνει πολιτική δουλειά για τη βελτίωση της κατάστασης γιατί οι γυμνία αριθμοί δίνουν μια διαφορετική εικόνα. 11,5 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Μόλις 500.000 ζώα λιγότερα από ότι το 2000. 8. Και έχουμε ήδη, ακόμα μάλλον χρησιμοποιούμε 7.000 πρωτεύοντα ζώα ακόμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τις, την εξέταση της κατάστασης. 32% των ε, ε, ουσιών που έχουν δοκιμαστεί σε πειράματα σε ζώτα ζώα κατά 92% όπως έλεγα απορρίπτονται μετά την πρώτη κλινική δοκιμή ενώ το 73% φαίνεται να δημιουργούν πολύ σοβαρές παρενέργειες παρά το ότι έχουν περάσει από τη δικασία του πειράματος σε ζώτα ζώα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι εναλλακτικέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κύτταρα, ιατρικό υλικό άλλου τύπου που μπορεί να αξιοποιηθεί Υπάρχουν ε, δηλαδή πρόοδοι τέτοιε οι οποίε μα επιτρέπουν να έχουμε εναλλακτικέ σε σχέση με τα πειράματα στον Ταζά. Μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε τι εναλλακτικέ αυτέ. και αν ναι, μπορούμε να δούμε τι είδου ε, διαδικασίε θα πρέπει να αντικαταστήσουν το κάθε τύπο πειράματο. Και μια ερώτηση για την οδηγία, περί λόγος. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί πλήρω αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει να κάνει και με την προστασία των ζώων εξασφαλίσει η προστασία των ζώων. Άρα πρέπει να βρούμε άλλου τύπου ε, νομοθέτημα που θα αντικαταστήσει το τμήμα που αφορά την προστασία των ζώων πριν καταργηθεί αυτή η οδηγία. Και κάτι ακόμη. Βλέπετε κάπου αλλού στον κόσμο εναλλακτικέ που να έχουν δοκιμαστεί και να είναι εφαρμόσιμες, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούνται ζώα ζώντα σε πειράματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Χάζεκαμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους ε, διοργανωτές της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ακούμε να εκφράζουν τη δυσφορία τους, την απόγνωσή τους πολλές φορές όλοι αυτοί οι ε, άνθρωποι που αντιδρούν τα πειράματα εις βάρος ζών των ζώων. Βέβαια, είναι γνωστό ότι δεν γίνονται σε συνθήκες διαφάνειας και έτσι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Αν είχαμε συνθήκες διαφάνειας σε σχέση με τα ε, πειράματα σε τα ζώα, θα είχαμε πολύ περισσότερες φωνές διαμαρτυρίας. 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε πειράματα σε εργαστήρια. Αλλά πολλά άλλα που βγαίνουν έξω από το βίντεο εφαρμογής της οδηγίας αντιμετωπίζουν κακομεταχείριση με αυτή την έννοια. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ζώα, με, με ζωντανά, με όντα τα οποία οφείλουμε να προστατεύουμε. Εάν διαπιστώνετε ότι είναι περιτές ή άχρηστες αυτές οι έρευνες που γίνονται με πειράματα πάνω στα ζωντά ζώα, απλούστατα πρέπει να σταματήσουν. Βλέπουμε να προβάλλονται κάποια επιχειρήματα τα οποία δεν αληθεύουν, ότι τα μπορούν τα πειράματα στα ζώα να προσφέρουν ε, περισσότερη ασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν αληθεύουν σε αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων στην ε, διαφάνεια των ε, πειραμάτων. Και θα ήθελα από τα τρία R που αναφέρθηκαν νωρίτερα, replacement, reduction and και refinement, δηλαδή αντικατάσταση, μείωση και ε, διευκρίνηση των όρων της ενέργειας ή της διαδικασίας, να έχουμε και το rehoming, δηλαδή τον επαναπατρισμό των ζώων όταν έχουν τελειώσει τα πειράματα. Και θα ήθελα να παρακαλούσα τώρα τον κύριο Τσούλο, λέει ο πρόεδρος, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους εισηγητές και ευχαριστώ τους οργανωτές για το, εξωτερικό το εξαιρετικό αποτέλεσμα του να συλλέξουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές για να γίνει συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πειράματα στα ζώα. Αυτό δείχνει την εμπλοκή των πολιτών στην καθημερινή πολιτική. Περνώντας τώρα στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της υποστήριξης της νέας μεθόδους πρόβλεψης μη χρήσης, μέσω μη χρήσης ζώων. Έχουν, έχει υπάρξει πρόοδος λόγω της επιστημονικής ακριβώς ανάπτυξης και υπάρχουν νέες διαδικασίες κύρωσης μεθόδων που δείχνουν ότι τα νέα συστήματα αυτά είναι αξιόπιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία πράγματι εξελίσσεται εδώ και αρκετό χρόνο, εδώ και δέκα περίπου χρόνια και δημιουργεί και αρκετά εμπόδια οικονομικά και γραφειοκρατικά. Αυτά τα εναλλακτικά συστήματα λοιπόν πρέπει να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν ζώα. Ε, πέρα από αυτό το πλεονέκτημα, μιας και είναι εγκεκριμένες μορφές συστημάτων, δεν πρέπει να περάσουν από νέες διαδικασίες επιστοποίησης. Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα, τα αποτελέσματά τους δεν ε, είναι εφαρμόσιμα στο ανθρώπινο είδος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν στρεβλωμένος ανταγωνισμός όπου αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι αντιμετωπίζουν τεχνητά εμπόδια. Ενώ οι μέθοδοι μέσω των ζώων έχουν εύκολη ζωή θα έλεγα. Γι' αυτό θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν θα προχωρήσει στην επανεξιολόγηση αυτών των συστημάτων πιστοποίησης έτσι ώστε οι νέες αυτές μέθοδοι να γίνουν ταχύτερες στην χρήση τους και να μην χρησιμοποιούν επιτέλους ζώα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροστά έχει το λόγο τώρα. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας να μιλήσω για την οδηγία 2010, την υπαριθμόν 63. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας την εξέθετησε, ε, παραθέτοντας επίσης το άρθρο 4 αυτής, το οποίο εξηγεί ότι οφείλουν τα κράτη-μέλη να κάνουν σεβαστούς τους όρους και να επαληθεύουν τους όρους ε, εφαρμογές της οδηγίας. Βεβαίως και εγώ μεριμνώ για την ευζοία των ζώων, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο της οδηγίας αυτής το οποίο προβλέπει δεοντολογικές ε, προϋποθέσεις υποχρεωτικές πριν ξεκινήσουν πειράματα εις βάρος των ζώων και βεβαίως υπάρχει Υπάρχουν και τα τρία R που αναφέραμε νωρίτερα, ε, το, η μείωση δηλαδή των πειραμάτων σε ζώτα ζώα, Δεύτερον, η αντικατάσταση ή μάλλον η χρήση τους, δηλαδή να μην γίνονται πειράματα σών εάν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και μόνο αν δεν υπάρχει εναλλακτική. Και τρίτον, η βελτίωση, δηλαδή η ως το δυνατόν πιο ε, βελτιωμένη χρήση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ της ευζοίας των ζώων και της ε, επιστημονικής ε, πρόοδου για να παραμείνει ε, στην ε, πρωτοκαθεδρία της βιοιατρικής έρευνας η Ευρώπη το 2017-2018 πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της ε, εφαρμογής της οδηγίας με βάση και τις πρόοδους της επιστήμης. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι προτιμότερο να γίνονται με σεβασμό των υψηλών προδιαγραφών σεβασμού των ζώων και της ψωίας τους τα πειράματα σε ζωντά ζώα παρά στον υπόλοιπο, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου που έχει χειρότερα επίπεδα προστασίας, διότι αν απαγορεύσουμε εμείς τα πειράματα στα ζώα, τότε αυτά θα γίνονται στην Ασία ή σε άλλες υπήρους, όπου δεν ισχύουν κανόνες προστασίας της ευζωίας των ζώων, όπου δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και θα ήθελα να επανέλθω για να ε, επιχειρηματολογής ορισμένων, εναντίον ορισμένων οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να ισχυριστούν ότι τα πειράματα σε ζώα μπορεί να θέτουν και σε κέντρο την υγεία την ίδια του ανθρώπου, του ασθενούς. Μα αντιθέτως η ε, οδηγία ίδια ορίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται ε, η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων. Δεν απαγορεύεται, δεν παρεμποδίζεται δηλαδή η αναζήτηση άλλων μεθόδων του αντίον, ενθαρρύνεται. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αναμφίβολα καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώς έχουν ξεκινήσει από πειράματα σε ζώα. Επί παραδείγματι, η μεταμόσχευση βλαστοκυτάρων καρδιάς, ε, η μέθοδος για την ε, μεταμόσχευση μετοχονδρίου ή η, η μέθοδος για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον έχουν γίνει έχουν αναπτυχθεί με βάση πειράματα που ξεκίνησαν από ζώα και ε, προηγμένα ζώα και ναι, έχουμε ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι, αυτοί οι πειρασματισμοί για να αναζητήσουμε τις εναλλακτικές και να συνεχίσουμε τις εναλλακτικές βεβαίως ε, από τα κύτταρα του ομφαλίου λόρου και τα βλαστοκύτταρα, να αναζητούμε βεβαίως εναλλακτικέ. Αλλά αν δεν υπάρχουν εναλλακτικέ θα πρέπει, δυστυχώς επαναλαμβάνω, να κάνουμε πειράματα σε ζώντα ζώα, έστω και αν αυτό δεν ευχαριστεί κανέναν και ιδίως αυτούς που εργάζονται στα εργαστήρια που είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν στα πειράματα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι η ερώτησή μου. Πώς εξηγείται όλες τις θεραπευτικές επιτυχίες που κατέστησαν δυνατές χάρη σε πειράματα σε ζώα, ζώντα ζώα, που μπόρεσαν να, έτσι να σώσουν ζωές, πώς είναι δυνατόν να απαγορευθούν. Βεβαίως και πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ. Βεβαίως, αλλά την οδηγία αυτή τη χρειαζόμαστε. Την οδηγία 2010 του 60, 63. Ε, e, bardzo proszę o ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ να αποφεύγετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και αντιδράσεις. Η κυρία Γκροστέτα ήταν, μίλησε εκ μέρους των Επιτροπών ΕΝΒΙΤΡΕ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Καπεθόνο Ρουής. Από τις επιτροπές επίσης αυτές και έχει το λόγιο δεκτά η κυρία Καπεθόνο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ καταρχάς να συγχαρώ όσους ε, με αυτή την άσκηση δημοκρατίας συμμετείχαν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι γιατρός και μελετώ ε, την επίπτωση που θα έχει η θεραπευτική αντιμετώπιση που συνιστώ κάθε φορά. Και έχω κάποια ερωτήματα. Πριν περάσω σε αυτό όμως να πω ότι όπως και στους περισσότερους νομίζω παρόντες, έτσι και σε μένα, δεν θα ήθελα να πρέπει να καταφύγω σε πειράματα ή δοκιμές σε ζώα για να πετύχω τη βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νόσων. Όμως δυστυχώς δεν είναι τόσο ανεπταγμένες άλλες ε, εναλλακτικές μέθοδοι ή δεν υπάρχουν καν ε, τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι. Μιλώ ιδίω ε, για τον αφιβληστοειδή ή ε, την in vitro, τις in vitro δοκιμές και πειράματα στον εγκέφαλο. Δεν γνωρίζουμε και θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδες μέθοδες. Έχουμε, μέθοδοι. Έχουμε πειραματικά μοντέλα, πληροφορικής ε, και άλλα που δείχνουν ότι υπάρχει πρόοδος αλλά με το Αλτσχάιμερ, το, την νόσο του Πάρκινσον και άλλες νόσες έχουμε μεγάλη πρόοδο χάρη και στα πειράματα σε ζωά. Μπορούμε έτσι να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους, να βελτιώσουμε την υγεία τους. Δεν μπορώ λοιπόν να, να πω ότι μπορούμε να καταργήσουμε σήμερα τα πειράματα σε ζώα, ούτε αυστηρό ε, και άκαμπτο τρόπο. Σίγουρα τα πειράματα αυτά βοήθησαν ε, στην ανάπτυξη πολλών εμβολίων για την αντιμετώπιση νόσων που μετά ήταν θανατηφόρες. Ε, επέτρεψαν την ανάπτυξη θεραπείων για σημαντικά στήματα, ινσουλίνη για τους διαβητικούς ε, και θα μπορούσα να παριθμίσω πολλές άλλες τέτοιες θεραπείες που ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων ασθενειών και από νομικής πλευράς να πω ότι τα πειράματα σε ζώα. Είπατε εσείς ότι δεν είναι απαραίτητα ή δεν είναι τα κατάλληλα γιατί δεν έχουμε την ίδια γενετική ταυτότητα άνθρωποι και ζώα. Όμως αυτό είναι μία φάση μόνο του πειραματισμού ε, για τη βελτίωση τη υγείας και την καταπολέμηση των ε, ασθενειών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε αυτή τη νομική πτυχή. Εάν μπορούσαμε να είχαμε παλιθέσει εκ των προτέρων η ταλιδομίδη τι επιπτώσεις ε, θα έχει στα ζώα. Σήμερα αυτή η ένωση ε, των ασθενών που διεκδικεί αυτά που διεκδικεί εδώ, να αναγνωριστούν δηλαδή αυτά τα καταστροφικά, ε, οι καταστροφικές βλάβες που προκαλεί αυτή η ουσία, δεν θα είχαν ξεκινήσει αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία. Άρα γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι προβλεπτικό μοντέλο. Επίσης, ξέρουμε ότι οι περισσότερες ε, θεραπείες προέρχονται από τέτοιες έρευνες, προέρχονται από τέτοια πειράματα. Άρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα με τη γενική ταυτότητα. Μακάρι 100% θα, να ήταν αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Όμως υπάρχουν επιτεύγματα και αυτά δεν μπορούμε να τα ε, δεν μπορούμε αυτό να το διαψεύσουμε. Για τους ε, πολίτες που λένε για την έρευνα στα ζώα το θέμα είναι ότι η θεραπεία ε, νόσων πολλές φορές δεν έχει να κάνει τίποτα με τη θεραπεία των νόσων, αλλά άλλοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν. Η οδηγία όπως υπόθηκε εδώ κατ' εμέ είναι καλύτερη που μπορούμε να έχουμε, είναι πλέον προηγμένη σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγγυάται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη και την καλή μεταχείριση των ζώων και μπορώ να σας πω ότι Σίγουρα ε, έχοντας ως βάση και αυτή την κριτική αναθεώρηση πιστεύω όμως ότι ο στόχο είναι, ναι μεν, να διασφαλίζουν τα κράτη-μέλη την σωστή εφαρμογή τη και αφετέρου να αναζητούν εναλλακτικέ μεθόδους. Δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι μπορούμε να αποκλείσουμε 100% σήμερα τα πειράματα και τις δοκιμέ σε ζώα. Δεν γίνεται. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους ε, διοργανώτες αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών, λέει ο κύριος Θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουν περάσει από θέματα ενδοκρινικών διαταρακτών και γενικά χρήση ε, των χημικών στην κοινωνία τελευταία πειράματα σε τα ζώα και μετά τον ειδικό ε, τρόπο δεξαγωγής των ε, πειραμάτων νομίζω ότι έχουμε μια σειρά από θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της οδηγίας του 2010. Έχουμε δηλαδή καταρχάς την δήλωση ότι αποφεύγουμε τα πειράματα σε ζώα και αλλά μια και εγώ έχω σπουδάσει βιοτεχνολογία και έχω κάνει και διδακτορικό, μπορούμε να συζητήσουμε Βρεταλάνθη και ε, αν θέλετε μετά να πιούμε ένα καφέ παρέα. Ε, για τον κύριο Γκίκ θα ήθελα να πω ότι η παρουσίαση του αποκλεί, η Γκρίκ θα ήθελα να πω ότι η παρουσίαση του αποκλεί οποιοδήποτε ε, προγνωστικό πρότυπο ή μοντέλο. Γιατί ούτε με, ανθρώπινη, με δοκιμές των άνθρωπων μπορεί να γίνει προγνωστικό μοντέλο. Άρα η αδίποτε ε, επιστημονική έρευνα μπαίνει στον πάγο. Α μιλήσω όμως και για την κυρία Γκροστέτ. Έχει γίνει πρόοδος στην επιστήμη, την ιατρική περίοδο, φαρμακευτική περίθαλψη και χάρη στο, στα πειράματα σε ζώα. Δεν είναι ικανοποιητικό αυτό. Πάντα πρέπει να κοιτάμε πώς λήφθησαν οι αποφάσεις. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να κοιτάμε να φτιάχνουμε και μοντέλα που θα εγκαταλείπουν το πρότυπο των ε, πειραμάτων σε ζώα, γιατί όλα αυτά τα μοντέλα στηρίζονται σε προηγούμενη έρευνα πάνω σε ζώα. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες των ναρκωτικών σε ε, ζώα ή μετά στον άνθρωπο. Πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα και νομίζω ότι η γνώμη της Επιτροπής έχει πολύ μεγάλη σημασία εφαρμόστε στα 28 κράτη-μέλη οδηγία, αλλά όχι με του ίδιου όρου και με την ίδια συνένεση. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο στη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τις ύψες τι προδιαγραφέ στον κόσμο για την έρευνα σε ζώα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα, στην ετροφαρμακευτική στη βελτίωση τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ε, για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Φαντάλ. Nie Αυτά και με Αποσιάζει από τη Ας ακούσουμε λοιπόν τους ειδικού μας. Α, όχι. Θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που έφτασα με τόση καθυστέρηση στη συνεδρίαση. Τρέχω από τη μια αίθουσα στην άλλη σήμερα. Είχα πολλέ συνεδρίασει. Θα ήθελα να πω δύο λόγια εκ μέρους των εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου και να ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις. Έχει υποστηρίξει τη σχετική οδηγία στο κόμμα των εργατικών της Βρετανίας γιατί θεωρεί ότι αποτελεί βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναζητούν εναλλακτικέ στις, ε, στο ιστορικό τους Τα τρία ρόλ λοιπόν αυτά, η μείωση, η, η αναλλακτικών και η βελτίωση των πειραμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα είχαμε υπογραμμίσει. Ιδιαίτερα λοιπόν είχαμε ζητήσει στόχους που όμως δεν περιελήφθησαν, στόχους ως προς τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν έχω την εξή ερώτηση, πολύ συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε δει και πολλά email από διαφορετικές θέσεις κάθε φορά και θέλω να αντιληφθώ ως Ευρωβουλευτής τι αλλακτική μπορώ να έχω σε σχέση με μια ε, διαδικασία πειράματος σε ζώντα ζώα ε, για σημαντικές ασθένειες όπως σε παραδείγμα τη σκλήρινση κατά πλάκας. Και τι μπορώ να κάνω σε εθνικό επίπεδο, στα κράτη-μέλη δηλαδή, ώστε οι αρχές αυτές της μείωσης εναλλακτικής κτλ. να εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη. Και σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τον ειδικό μας τον κύριο Greek. Ναι, θα προσπαθήσω σήμερα τώρα να μην ε, ξεπεράσω το χρόνο μου. Δεν θα ήταν λογικό φυσικά να περιμένω ότι θα αντιληφθείτε πλήρως όλοι σας όλα τα επιστημονικά δεδομένα με τα οποία σας κατέκλυσα σήμερα. Ε, έχω μελετήσει πάρα πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Ελάχιστοι είναι οι επιστήμονες που αντιλαμβάνονται την επιχειρηματολογία μου. Η κοινωνία όμως ενολοπλήτεται άμεσα και έμεσα από τα πρότυπα αυτά. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει με σοβαρότητα να σώσει τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που κινδυνεύουν από ασθένειε τύπου νευρολογικού φερρυπίν, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πιο αποτελεσματικά μπορεί και να αξιολογήσει την πρωτοβουλία αυτή κατά τρόπο θετικό. Και εκείνοι οι οποίοι προσπίζονται τα μοντέλα των πειραμάτων σε ζώα, αλλά και ο υποφαινόμενος. Πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο να παρουσιάσουμε τις επιχειρηματολογίες μας και να απαντήσουμε διεξοδικά σε όλα τα ζητήματα τα οποία ηγέρθησαν σήμερα. Εγώ εδώ και καιρό ήθελα να το κάνω. Αλλά η κοινότητα η οποία υποστηρίζει ε, τα πειράματα εις βάρος ε, των ζώων δεν επιτρέπει τις ευκαιρίες και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ εύγλωτο. Εγώ θα ήθελα να γίνει συζήτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να διαθέσω στο δυνατό χρόνο. Θέλω οι ειδικοί για τα θέματα αυτά της επιστήμης να είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν τις θέσεις μου. Και μετά μόνο να γίνει συζήτηση. Και τα επιχειρήματα. Και επίσης παρακαλώ, πείτε μου, ακούσατε επιχειρήματα σήμερα. Είναι όλα αυτά ισχυρισμοί. Είναι ισχυρισμοί ότι έχει γίνει αυτό και εκείνο και το άλλο με επιτυχή τρόπο χάρη στα πειράματα. Και εγώ μπορώ να ισχυριστώ λοιπόν ότι έχω πάει στο φεγγάρι και έχω γυρίσει και έχω δουλέψει κιόλας εκεί. Ε, δεν έχω δουλέψει όμως στο φεγγάρι. Ο επιστήμονας έχει ένα ιστορικό καθήκον. Κάθε φορά που έχω κάνει την έρευνά μου για το πού έγιναν οι δεξεκέλευτες ανακαλύψεις, τα πειράματα στα ζώα δεν είχαν παρά μηδανικό ή και καθόλου ρόλο να διαδραματίσουν στις μεγάλες αλλαγές στην ιατρική περίθαλψη. Και μάλιστα πολλές φορές παρουσιάστηκε ρόλος ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Για την ε, σύγχρονη πολιομιελίτιδα, την HID, θα είχε ανακαλυφθεί το εμβόλιο 40 χρόνια νωρίτερα εάν δεν είχαν γίνει παραπλανητικά για τους, ιστορι... για τους ιατρούς πειράματα σε πυθίκους. Και έχω εκατοντάδες άλλα παραδείγματα να σας δώσω. Μην πιστεύετε λοιπόν αυτά που σας λένε, μην πιστεύετε ούτε εμένα. Να κάτσουμε δύο-τρεις εβδομάδε να δώσουμε το χρόνο να γίνει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση ώστε εσείς οι ευρωβουλευτές, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσετε να λάβετε απόφαση με τα λόγου γνώσεως. Bardzo Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλει ο να λάβει το λόγο. Όχι. Καλώς τότε. Ας ακούσουμε τους ε, ε, πρωτοβουλίας. Ο κύριος Μενάς πρώτα. Ο χειρός κτηνίατρος λέω στον κόσμο ότι εγώ δεν θα ήθελα ένα φάρμακο για τα άλογα να το δοκιμάσω σε ένα παπαγάλο και γελάνε ε, αυτοί του οποίους γιατί καταλαβαίνουν αμέσω ε, το μήνυμα. Αν δεν θέλουμε τα φάρμακα που προορίζονται για άλογα να τα δοκιμάσουμε σε παπαγάλους, γιατί θέλουμε φάρμακα που προορίζονται να τα δοκιμάσουμε σε ζώα. Είναι πολύ λογικό αυτό το επιχείρημα. Είμαι μέλος δύο επιτροπών διοντολογίας και ηθικής για τα ε, ζώα, την κρατική των ζώων και πραγματικά με απογοητεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν μπορώ ε, να προσβάλλω την εγκαιρότητα του ζωικού μοντέλου. Μου λένε ότι πρέπει να επιμείνω σε αυτά τα τρία άρα, αντικατάσταση, μείωση, βελτίωση που αναφέρονται στην οδηγία και δεν μπορώ να υπερβώ αυτά τα όρια, τα όρια που θέτουν αυτά τα τριάρια, επομένω δεν μπορώ να προσβάλλω την εγκυρότητα του ζωικού μοντέλου. Σήμερα μεγάλο μέρος τη έρευνα γίνεται σε ποντικούς, έχει να κάνει με την αντικαρκυνική έρευνα. Και ε, οι ζωικοί έρευνες θα πούνε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυτάρων και πολύ σωστά τα λέει αυτά ένα ερευνητή, γιατί δεν μπορεί το νοσοποιητικό σύστημα ενό ποντικού να το μελετήσει κανεί ε, σε καλλιέργεια άνθρωπων κυτάρων. Θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθεια στο να κάνουμε ε, έρευνα, ενώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την τεχνολογία με την, για τη χρήση ανθρώπινων δεδομένων, τον των άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν δεν ε, κατάφερε να αμφισβητήσει την επιστημονική εγκυρότητα των ζωικών πειραμάτων ή οδηγία ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία, γιατί σχεδόν όλη η έρευνα και οι προτάσει ε, για την έρευνα στα ζώα αιτιολογούνται με το ότι να ορίστε τι θα κάνω σε ένα ποντικό και ίσως έτσι βρω θεραπεία για και μετά βάλτε ό,τι θέλετε. Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, καρκίνο, σκλήρωση καταπλά... καταπλάκες και το καθεξής. Στη βιβλιογραφία την επιστημονική βλέπουμε ότι οι ε, πιθανότητες της ε, βασικής έρευνας, ε, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση. Μπορεί να σα πούνε οι ζωοκινητικέ, ναι, όχι, έχει εφαρμογή σε ανθρώπινε νόσου. Όχι. Όλη όμω η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι πιθανότητε, η βασική έρευνα να οδηγήσει σε ένα κλινικό αποτέλεσμα είναι τη τάξη του 0,004%. 0,004%. Επομένως θα πρέπει να διερωτώμαστε, είναι αυτός ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να χρησιμοποιούμε τους πόρους, ε, τα χρήματά μας ε, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η απάντηση είναι καταφατική. Και επαναλαμβάνω ότι η οδηγία ουσιαστικά πρόδωσε και την εμπιστοσύνη τη κοινή γνώμη ό,τι αφορά τη σύνθεση επιτροπών διοντολογία και ηθική, ε, που ουσιαστικά έκλεινε ε, υπέρ ε, τη έρευνα έρευνας ζώα. Και δεν προώθησε τι αναλυτικέ μεθόδου. Ούτε είχε σε, αυτή, σε επιτροπέ, υπήρχαν, προσωπούνταν αρκετά ε, υπέρ των, των εναλλακτικών μεθόδων. Αν προσπαθούμε να προσβάλλουμε εντό αγωγικών έναν ερευνητή ζωικό λέγοντας ότι θα πρέπει να κάνει ε, κάτι που σχετικά με, με, με τους ανθρώπους. Θα πρέπει να βρει μάρτυρες, θα πρέπει να βρει δικηγόρους κτλ. Είναι δεμένα τα χέρια μας, ε, διότι έχουν και την πίτα και την τρώνε όσοι κάνουν έργα στα ζώα. Bardzo dziękuję. W ten sposób zamknęliśmy pan. ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο κομμάτι των συζητήσεών μας και ευχαριστώ τους ειδικούς μας. Θα παρακαλέσω τώρα τους, ε, τον καθηγητή, την καθηγήτρια Μπαρέσινου έρθει εδώ και σαν σχόλιο θα ήθελα να πω το εξής. Όλους μας μας ενδιαφέρουν τόσο και η ευζοία τους. Η μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο είχε σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, πώς αντιδρά και πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε ε, ασθένειες. Μπορούμε ίσως τώρα πια να μιλούμε για ε, θεραπευτικές μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως είμαστε υπέρ τέτοιων εξελίξεων όλοι μας. Αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε τις πρακτικές πτυχές ή ασδήποτε έρευνας μπορεί να διεξαχθεί χωρίς πειράματα σε ζώα. Δηλαδή, τι είδους επιστημονική βάση θα έχουν οι έρευνες αυτές. Ε, περιμένουμε την κυρία καθηγήτρια να λάβει το λόγο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που την βλέπουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Η παρουσία της βεβαίως είναι πολύτιμη για την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση καταρχάς. Αναλαμβάνω λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Καταρχά, να συμμετάσχω σε αυτή τη δημοσιακή ακρόαση και να ανταλλάξουμε απόψει ε, σε ό,τι αφορά την έρευνα στα ζώα. Συμπληρωματική σε πολλά άλλα μοντέλα που έχουμε σήμερα. Όπως προελέχθη, η έρευνα πρέπει να γίνεται από την κούνια μέχρι την κλίνη του εργαστηρίου και να επανέρχεται, αν θέλετε, μετά στην κούνια. Αυτό μπορεί να υπόθηκε με 30 χρόνια, αλλά υπάρχει και κάτι ε, που λείπει. Και ο κύριος Μπρένερ που το είπε αυτό δεν νομίζω ότι θα είχε αντίρρηση να προσθέσουμε τα μοντέλα σε αυτή την ε, πορεία. Γιατί λοιπόν τα ζωικά μοντέλα είναι για την έρευνα και στον άνθρωπο και στα ζώα θα έλεγα γιατί όπως υπόθηκε προηγουμένως σίγουρα υπάρχουν γενετικές διαφορές μεταξύ ζώων και κατά την, απο... κατά την ε, μάλλον από τις γνώσεις μου, το 90% ε, είναι ταυτόσημα, αλλά ποτέ 100% βέβαια, αλλά υπάρχει 1% ταύτιση. Και οι άνθρωποι και άλλα φυλαστικά έχουμε τους ίδιους ιστούς, τα ίδια όργανα, η φυσιολογία ομοιάζει πάρα πολύ. Αναφέρθηκε επίσης ότι πολλές ασθένειες είναι κοινέ για τον άνθρωπο και για διάφορα είδη ζώων, ο διαβήτης, ο καρκίνος, ανοσολογικές νόσεις, νόσεις που πλήττουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και πολλές άλλες λοιμώξεις, ε, όπως μεταξύ αυτών και το AIDS. Δεν υπόθηκε όμως ότι στο 90% το 90% των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι τα ίδια ή πάρα πολύ όμοια με αυτό το οποίο αναπτύσσονται για, την, ε, για τον άνθρωπο. Γιατί είναι πολύτιμα τα ζωικά μοντέλα ε, και για την έρευνα στα ζωή και για την έρευνα στον άνθρωπο. Φυσικά πρόκειται για μοντέλα. Δεν περιμένει κανείς ένα μοντέλο να είναι ταυτόσιμο με ένα άλλο. Δεν είναι τα ζωικά μοντέλα ταυτόσιμα με ε, τον άνθρωπο, ούτε το ένα είδος με ένα άλλο. Υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές αυτές, ε, να σας πω εν παρόδο, πρέπει να ληφθούν υπόψη με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά οι διαφορές τους είναι πολύ λιγότερες από τις ομοιότητές τους. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνούμε και υπόθηκε και αυτό. Έχουμε μεγάλη πολυμορφία στους ανθρώπους και διαφορετικότητα. Και αυτό εξηγεί γιατί πολλές φορές αντιδρούν ή ανταποκρίνονται πολύ διαφορετικά οι άνθρωποι στις διάφορες νόσους, αλλά ή στο ίδιο εμβόλιο ή στο ίδιο φάρμακο. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και στα ζώα. Ακριβώς λόγω της διαφορετικότητας, πολυμορφίας των ζώων. Βέβαια τα ζωικά μοντέλα σίγουρα χρήζουν βελτίωσης και έχουν βελτιωθεί ήδη με την πάροδο των ετών λόγω της επιστημονικής πρόοδου. Και μοιάζουν όλο και περισσότερο με τις ανθρώπινες ασθένειες. Έχουμε μη επεμβατικές τεχνικές όπως είναι οι τομογραφίες για παράδειγμα, οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ε, μελέτη ζωικών μοντέλων. Πολλά ε, επιτεύγματα μπορούμε να καταγράψουμε λόγω των ζωικών μοντέλων. Δεν θα σας τα απαριθμίσω όλα. Άλλοι μίλησαν για το διαβήτη για παράδειγμα. Εμβόλια. Για την πολιομήλυτα βέβαια ακούσαμε ότι το εμβόλιο για την πολιομήλικτα ή για την υπατήτηδα. Εγώ νομίζω ότι αποδείχθηκε η δράση τους σε ζώα πρώτα απ' όλα, σε ζωικά μας. Δύο με τρία εκατομμύρια ε, θανάτους αποφεύγουμε ε, το χρόνο χάρη στα εμβόλια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα στα εμβόλια. Αναφέρθηκε ο ιός του AIDS. Και πρέπει να πω, είμαι μία ε, γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά τι έχει συμβεί ε, στον τομέα αυτό ήδη από τη δεκαετία του 80. Και πολύ σωστά λέτε ότι τα δεδομένα δεν ήταν πολύ πτυχμένα. Μιλήσετε για 100 εμβόλια. Ε, δεν με ενδιαφέρει το νούμερο εμένα βέβαια. Ακόμη και αν κάποια φάνηκε να είναι αποτελεσματικά σε μοντέλα ε, πυθίκων, ε, σε ανθρώπους δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Γιατί φταίει το μοντέλο του ζώου, το ζωικό μοντέλο ή ο επιστήμονας, η επιστήμη. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αν κανείς δει καλά το πείραμα, παραδείγματος χάρη για την έρευνα συμβόλου κατά του AIDS, Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή δεν χρησιμοποιούσαμε το σωστό μοντέλο, δεν χρησιμοποιούσαμε ε, το, σωστούς, ε, το σωστό ιό, δεν χρησιμοποιούσαμε ούτε το σωστό σημείο εμβολιασμού, ούτε είχαμε θέσει ουσιαστικά τα σωστά ερωτήματα για να έχουμε σωστή απάντηση. Ο τομέας αυτός πάντως σήμερα παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Χρησιμοποιούμε κάποια αντισώματα τώρα, τα οποία έχουν αναπτύξει οι επιστήμονες. Και αποδείχθηκαν ήδη σε ζωικά μοντέλα ότι είναι αποτελεσματικά για τη μείωση του μεγέθους του λεγόμενης δεξαμενής για τον HIV. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν μπορεί να σταματήσει την θεραπεία ένας ασθενής. Σίγουρα ξέρουμε όμως ότι με αυτό το μειώνεται η δεξαμενή αυτή και τα βεβαιώσαμε πέραν των ζωικών μοντέλων αυτά τα στοιχεία και στον άνθρωπο. Αυτό για να σας πω ότι χρειαζόμαστε τα ζωικά μοντέλα ακόμη και αν έχουν τα ωριά τους. Όπως τα άλλα μοντέλα, εναλλακτικά. Και αυτά έχουν τα δικά τους όρια. Οι εναλλακτικές μέθοδοι που έχουμε σήμερα είναι στο ε, οι δοκιμέ στο Σολίνα, ε, οι ε, τα υπολογιστικά μοντέλα και άλλα. Βελτιώνονται τεχνικές από τους ειδικού. Σας πω ότι στη χώρα μου τη Γαλλία το 80% των ερευνητών που χρησιμοποιούν ζωικά μοντέλ ξεκίνησαν με ε, μια εναλλακτική μέθοδο. Και μόνο όταν δεν έχουν άλλη επιλογή συνεχίζουν να συλλέγουν δεδομένα. Τα οποία είτε επιβεβαιώνται είτε όχι. Από την αλληλεπτική μέθοδο. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα εναλλακτικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί δεν μπορούν να καλύψουν τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ιστών και των οργάνων που υπάρχουν στον οργανισμό. Άρα πρέπει στο μέλλον να αναπτύξουμε καλύτερε αναλυτικέ μεθόδου και σίγουρα είμαστε θετικοί ότι θα έχουμε τέτοια πρόοδο στο μέλλον. Τα ζωικά μοντέλα βέβαια από μόνα του δεν είναι επαρκή για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Πρέπει να περάσουμε και σε κλινικέ μελέτε στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικέ οι μελέτες στου ασθενεί. Στον τομέα το δικό μου, τον τομέα του AIDS, και αυτό νομίζω έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν για τη γενετική. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς ε, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί, έχουν αντοχή ε, στην ε, προσβολή από τον ιό του AIDS. Είναι λιγότερο από το 3% αλλά αντιστέκονται και δεν μονοσούν αυτό το 3%. Και από αυτό έχουμε εκπονήσει κάποια ζωικά με το οποίο είναι πολύ αντιπροσωπευτικά των αντιποτελεσμάτων που παρατήρησαμε στον άνθρωπο. Δεν έχουμε την επιλογή όμως, δυστυχώς, εάν θέλουμε να απαντήσουμε ορισμένα από τα ερωτήματα και κάποια από αυτά γύρονται από την παρατήρηση των ασθενών, θα πρέπει να πάμε στις αλληλικές μεθόδους, να ζητήσουμε ε, απαντήσεις από τα ζωικά μοντέλα και να επανέλθουμε στις κλινικές δοκιμές με τους ασθενείς για να ε, επικυρώσουμε ή όχι τις υποθέσεις μας αλλά και τα αποτελέσματα και στο σωλήνα, και in vivo και in vitro τέλος πάντων. Ολοκληρώνοντας για τα 3R πιστεύω ότι με την οδηγία αποκνόμεσα στην ανάγκη να προστατεύσουμε τα ζώα και τον άνθρωπο και χρειαζόμαστε την έρευνα στα ζώα αν θέλουμε να συνεχίσουμε, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και την υγεία τους. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω και το έχω πει και κατά το παρελθόν ότι ο κανονισμός για το ζεκαμαντέ είναι παρόμοιος, δεν μοιάζει 100% στον κανονισμό περιφυκής και το λύζει τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Και ολοκληρώνω με ένα παράπονο κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε ασθενείς εδώ για να πούν και αυτή την άποψή τους. Αυτό έτσι λίγο με λυπεί. Και επειδή έχω βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ, πρέπει να πω ότι επειδή έκτοτε με επισκέφθηκαν πολλοί ασθενεί, ε, θέλω να είμαι η φωνή τους και αυτό προσπαθώ σήμερα, να είμαι η φωνή αυτών των ασθενών. Είμαι βέβαια ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσουμε την έρευνα στα ζώα σήμερα, αυτό θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή και για την υγεία των ζώων και για την υγεία του ανθρώπου. Να έχετε υπόψη ότι το καθήκον μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ασθενών. Και έχουμε το χρέος να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή αλλά και τη ζωή του ζώου. Και νομίζω ότι όλοι εδώ σήμερα ουσιαστικά συμμεριζόμαστε αυτή την ιδέα. Και ολοκληρώνω με μια ενθάρρυνση που θέλω θα ήθελα να ενθάρρυνω την ευρωπαϊκή κοινότητα να στηρίξει περισσότερη έρευνα σε εναλλακτικέ μεθόδους για το μέλλον, για να μπορέσουμε να αποκριθούμε στις ανάγκες. Νομίζω ότι όλοι με πολύ μεγάλη χαρά θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγήτρια για την έξοχη αυτή δήλωση. Και πάνω απ' όλα την επισήμανση ότι πρέπει να λάβει υπόψη και οι προσδοκίες των ασθενών. Ας περάσουμε τώρα στο γύρο των έρωτα αποκρίσεων. Ο κύριος Ταραμπελά πρώτος για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πολλοί ομιλητέ είπαν αυτά που θα ήθελα να πω. Σεβόμεθα τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών. Σωστός ο στόχος. Λιγότερες δοκιμές με ζώα. Λιγότερη δυστυχία για τα ζώα. Είμαστε σε μια παρακμιακή βέβαια πολιτιστική κατάσταση γιατί οι δηλώσεις για την ευημερία των ζώων είναι πολύ περισσότερες από την πείνα στον κόσμο ή από τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες. Εν περιπτώσει πρέπει να σεβαστούμε όμως αυτήν την πρωτοβουλία των πολιτών. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κάμπεσον Ρουίζ όπως επίσης και με την κυρία Γκροστέτ λέγοντας ότι έχουμε προσπαθήσει εμείς να μειώσουμε ε, τις δοκιμές αυτές. Το να πούμε όμως αμέσως σταματήστε τη χρήση των ζώων αυτό θα ήταν εγκληματικό. Έχει υπάρξει πρόοδος σε κάποιους τομείς. Σε έναν κόσμο χημικό και εμολυσμένο έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Ένα χρόνο κάθε τέσσερα χρόνια ίσως σε κάποια φάση να σταθεροποιηθεί χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και χάρη στα πειράματα με ζώα. Φυσικά και πρέπει να ακούσουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες και να τα συνδυάσουμε με την κοινωνική ευημερία. Μια πρωτοβουλία σαν παράδειγμα για την αποκατάσταση της ε, θανατική ποινή όπως ο κύριος Όρμπαν στην Ουγγαρία. Θα υπάρξουν εκατομμύρια. Οι πολιτικοί θα πρέπει να υπακούσουν σε αυτό. Όχι, θα πρέπει μερικές φορές να είμαστε αντίθετοι με το ρεύμα. Και τελειώνω πρόεδρε. Ο, να πω ότι η δήλωση αυτή ε, απαιτεί σεβασμό. Οι ε, επιστήμονες που είναι εδώ θα πρέπει να τους ακούμε φυσικά, αλλά οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν τις απαιτούμενες διαιτησίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Κυρία Χόιμπουχ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι πράσινοι είχαν καταψηφίσει το 2010 την οδηγία αυτή, διότι θεωρούμε ότι η προστασία των ζώων και η απέτηση για ε, προώθηση μεθόδων χωρίς πειράματα σε ζώα δεν εξασφαλίζονταν τον αντίον, σε μας περιπτώσεις επιδεινώθηκε η κατάσταση. Και βεβαίως, ε, σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι έχουμε υποδειγματική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλω να επισημάνω τα κράτη-μέλη, το καθένα χωριστά, δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουν και να επιβάλλουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις από αυτή την οδηγία. Τεράστια έλλειψη. Και διαρωτώ με γιατί έχει επιβληθεί αυτή η απαγόρευση. Τα ζώα υποφέρουν για να υποβληθούν σε δοκιμές που δεν μεταφέρονται στον άνθρωπο αυτές καθεαυτές. Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές σε ζώα, σε πειράματα, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν για φάρμακα. Κλασικό είναι το παράδειγμα του έρευνας για το AIDS, όπου ξοδεύτηκε πολύς χρόνος και χρήμα και κόπος από τη δεκαετία του χωρίς να έχουμε φτάσει ύστερα από 200 εμβόλια για το ζώα, δεν έχουμε εξασφαλίσει ούτε ένα για τον άνθρωπο. Έχουμε επίσης για να μελετήσουμε τις γενετικές μεθόδους τροποποίησης κάνει πειράματα σε ζώα που προξενούν μεταλλάξεις, οι οποίες στη συνέχεια καλύπτονται με διπλώματα εύρεσης τεχνίας. Και έτσι φέρνουν περισσότερο χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι τα πειράματα όχι μόνο δεν τείνουν να μειωθούν, αλλά θα ενισχύονται συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια μέθοδο χωρίς πειράματα σε ζώα για να μπορούμε να μεταφέρουμε και ε, λύσεις ε, ερευνητικές και διαδικασίες ερευνητικές οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται και να εφαρμόζονται στον άνθρωπο. Ξέρετε βεβαίως όταν μας λέτε ότι οι ασθενείς σας, ζητούν να υποστηρίξετε τα πειράματα σε ζώα, ξέρετε πολύ καλά ότι οτιδήποτε έχει γίνει στο χώρο της ευζοίας των ζώων και της απαγόρευσης των περιορισμών των πειραμάτων οφείλεται στις αντιδράσεις και τις γνώμες και κυρίως στην περίπτωση των καλλιντικών τα οποία χρησιμοποιούνταν πάνω σε ζώα χωρίς άλλο σκοπό παρά μόνο την παραγωγή καλλιντικών προϊόντων. Ε, ε, Κυρία Σάντρα Ροντρίγκε, καταρχά θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία που μα δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε αυτό το διάλογο. Επίση θέλω να πω ότι δεν είμαι ειδική για το θέμα αυτό που συζητάμε, όμω νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστούν όλες οι απόψεις, ε, όλες οι επιστημονικές γνώσεις, ε, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τις αποφάσεις ε, και σε προσωπικό επίπεδο καθένα αν θα κληθούμε να αποφασίσουμε πώς προσέχουμε την υγεία μας ή όταν είμαστε μέλη φορέων οργάνων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία αυτή τι στόχο έχει. Να δούμε κατά πόσον η χρήση πειραμάτων ε, στα ζώα είναι χρήσιμη ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια ευρεία συζήτηση, να έχω μια ροή πληροφοριών και σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί πάντοτε Έχουμε τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μεγάλα εργαστήρια, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους ομίλους, φαρμακοβιομηχανίες, αλλά όχι τόσο ε, άλλες επιστημονικές γνώσεις ή πρόσβαση σε άλλους φορείς, που εμένα όμως θα με ενδιαφέρει περισσότερο. Και νομίζω ότι και τους πολίτες, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές χρειάζεται να εφαρμόσουμε και την κοινή λογική. Τούτου λεχθέντος, έχω ένα ερώτημα. Υπάρχει σχέση μεταξύ του είδους της έρευνας που διεξάγεται με τα ζώα και το ότι σήμερα τρίτη αιτία θανάτων στον κόσμο είναι τα φάρμακα. Κυρία Γκαρδίνη, παρακαλώ. Hello, I replaced Madame Gardini. Αντικαθιστώ την κυρία Γκαρδίνη. Δεν είμαι η κυρία Γκαρδίνη. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Μπουσόη. Σέβομαι την πρωτοβουλία των πολιτών. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άκουσα και τις παρατηρήσεις της κυρίας Μπαρέ συνουσή και νομίζω ότι η επιστημονική πρόοδος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομακτική πρόοδο. Η οδηγία των τριών R αγγλικών είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η πλήρης κατάργηση της χρήσης των ζώων θα οδηγήσει τους ερευνητές εκτός Ευρώπης. Η έρευνα σε ζώα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση των ασθενειών. Εγώ πήρα μέρος σε δύο workshop τους τελευταίους μήνες, στην τελευταία συνάντηση ήταν οι υποψήφοι ή μάλλον αυτοί που κέρδισαν το Νόμπελ φαρμακευτικής το 2014 και είπαν ότι αν δεν είχαν τις δοκιμές σε ζώα στη διάθεσή τους δεν θα έπαιρναν ποτέ το βραβείο. Για την βιοιατρική έρευνα λοιπόν είναι απαραίτητη η χρήση των ζώων και έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλύτερη αντιμετώπιση ασθενειών όπως των καρδιολογικών προβλημάτων των γυναικών όπου έχουν υπάρξει πολλά βήματα. Παρά τις τελευταίες εξελίξεις για τις εναλλακτικές μεθόδους όπως τα ανθρώπινα κύτταρα και τα ανθρώπινα πρότυπα ε, ακόμα οι μέθοδοι αυτοί δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν πλήρως την χρήση των ζώων. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι για πορελς ασθένειες, περίπλοκες ασθένειες θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας έναν ε, λειτουργούντα ε, ζωντανό οργανισμό. Μιλήσατε εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο κύριος Σάικ επίσης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση και γι' αυτό θα ήθελα να ε, θέσω ε, ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο δεν έχει καλυφθεί στη συζήτηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε την τρίτη πρωτοβουλία πολιτών με ένα 1,1 εκατομμύρια πολίτες από 26 κράτη-μέλη που υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία με την υπογραφή τους. 80% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απορρίψει την, ε, ε, τον πειρασματισμό σε ζώντα ζώα γιατί δεν δέχονται να φωνεύονται ζώα και δεν δέχονται τις ε, φρούδες υποσχέσεις ότι θα μειωθούν τα πειράματα σε ζώα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να θεωρούνται τα ζώα ως μονάδες παραγωγής ούτε ως χρήσιμα μοντέλα οι αδίποτε πειράματα. Αυτή την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να τη υπόψη. Εάν ναι, όμω αποφασίσει το αντίθετο θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα απώλεια εμπιστοσύνη από τον πολίτη και το χάσμα, το κενό ανάμεσα στον πολίτη και τα θεσμικά όργανα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Θα είναι δε πολύ πιο δύσκολο στο μέλλον να μιλούμε για ιδεώδη, για ε, κοινωνία αξιών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε εδώ Εάν η πολιτική δεν το πράξουν, προφανώς θα πρέπει και να μας ε, ε, κάνει να απορούμε που χάνεται η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, την πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία 2000 του 1963 έλεγε ότι θα πρέπει να μην γίνονται πείραματα σε ζώνη εφόσον δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Αλλά δεν μπορούμε να λησμονούμε τι σημαίνει πόνος για τα ζώα. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Πρέπει να πούμε όλοι όχι στα πειράματα και πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές μεθόδους. Η οδηγία του 2010 δεν είναι καλύτερη. Διαφορετικά δεν θα είχαμε κάθε χρόνο 12 εκατομμύρια πειράματα σε ζώντα ζώα. Το καλύτερο της οδηγίας αυτής όμως είναι ότι βοηθά τις ατροφαρμακευτικές βιομηχανίες βοηθάει αυτούς που κάνουν πειράματα. Δεν βοηθάει όμως τον άνθρωπο και τις λύσεις για τους γιατρούς. Γι' αυτό πρέπει να αναστηθούν εναλλακτικέ μέθοδοι. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω τον στόχο της αντικατάστασης ε, της χρήσης των ζώων με εναλλακτικές στρατηγικές που να είναι άμεσα σχετικές με το ανθρώπινο όν. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν νομίζω ότι η προσωρινή αναβολή ισχύω τη συγκεκριμένη οδηγία είναι απαραίτητα ο καλύτερο ή ο μοναδικό τρόπο. Θα συμφωνήσω με την κυρία Μπαρέ Σινουσή για το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να προχωρούμε σε διαβουλεύσεις σε επιστημονικό επίπεδο χωρίς να εξαρτηθούμε αποκλειστικά σε πειράματα σε ζώα. Ένα μεγάλο τμήμα της ιατρικής έρευνας βασίζεται σε κάποια αναπαραγωγή των συμπτωμάτων των ανθρώπων σε άλλα ζώα. Τα, ενώ πάρα πολλοί γιατροί διαφωνούν τελικά με τη μέθοδο αυτή. Μία μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας έδειξε ότι το 95% των φαρμάκων τα οποία φαίνονται ασφαλή και αποτελεσματικά στα ζώα απέτυχαν την, τον κλινικό έλεγχο στους ανθρώπους λόγω απρόβλεπτων τοξικών συνεπειών στους ανθρώπους και λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα των ανθρώπινων ασθενειών, των ανθρώπων όσων, χωρίς ε, να προσπαθούμε να μιμηθούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά σε άλλα είδη. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί ε, την βασική αρχή της πλήρους ε, ακύρωσης των πειραμάτων στα ζώα και να δεχθεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας όπως επίσης και της Ανθρωπιστικής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρξει αναθεώρηση ε, της κοινοτικής νομοθεσίας όπου αυτό χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε εξ ονόματος της Επιτροπής ΣΥΤΡΑ από όπου και η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κύριε Σύνουση και κάθε σεβασμό προς την συμβολή της στην επιστήμη. Στο παγκόσμιο επίπεδο. Είμαι νέα βουλευτή, δεν συμμετείχα στη διαπραγματεύση τη οδηγία του 10. Ω καινούρια λοιπόν για αυτά τα θέματα, αλλά είμαι και μέλο Επιτροπή Ήτρε, που είναι αρμόδια για τα ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω στο άξονα τον επιστημονικό. Τα ηθικά, την ηθική συζήτηση την αφήνω για άλλους. Θα είχα λοιπόν τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον, μετά την ανακλέψη του ΕΣΤΟ το 1983, αφιερώσατε ένα μέρος της έρευνάς σας στην ανάπτυξη ενός εμβολίου. Θα ήταν δυνατή σήμερα η έρευνα αυτή χωρίς ε, πειράματα σε ζώα και χάρη στις τεχνολογίες. Δεύτερο ερώτημα. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων που είχατε στα ζώα, μεταφορά των αποτελεσμάτων στον άνθρωπο. Τρίτον, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επανεξετάζει την νομοθεσία και ας πούμε ότι απαγορεύει τα πειράματα σας. Αυτό τι ε, αντίκτυπο θα είχε στη δική, στη δική ερευνητική δουλειά. Και κυρίως ό,τι αφορά την αναζήτηση ενό συμβολίου για την αντιμετώπιση του AIDS και του, του έμπολα, γιατί όχι. Και τελευταίο ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα εργαλείο ερευνητικό, πάρα πολύ σημαντικό, που είναι ορίζοντα 2020. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε αυτό το ερευνητικό εργαλείο να το χρησιμοποιήσουμε για να αναζητήσουμε εναλλακτικέ μεθόδους αντί των πειραμάτων στα ζώα. Pan poseł Becker. Bakel. De Bakel. Bardzo proszę, bardzo proszę. Thank you, Chair. Um... Κύριος Δεμπάκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι σαφή νομίζω οι θέσει των διαφορών ομάδων, όπω υπόθηκαν μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να γίνει λογική συζήτηση και συμφωνώ με τον κύριο Ταραμπέλο ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο η επικράτηση της πλειονοψηφίας ή η τυραννία της πλειονοψηφίας. Πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε και την άλλη όψη και τις θέσεις της άλλης πλευράς. Από αυτούς που μίλησαν σήμερα λοιπόν και κυρίως από τους επιστήμονες καθίσταται σαφές για μένα το γεγονό ότι παρότι υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, και ανεπάρκειες ε, στο χώρο της έρευνας και από τα στοιχεία που δίνονται υπάρχουν βέβαια οι ανεπάρκειες αλλά πάνω απ' όλα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο Έχουμε μειώσει στο ίμιση ήδη ε, τα πειράματα. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι είναι καλύτερη η Ευρώπη με ή χωρίς πειράματα. Για μένα η απάντηση είναι θετική. Ε, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο και υπάρχει η απαντηση ειναι θετικη εχουμε κανει σημαντικη προοδο και υπαρχει η αντικατασταση τα διαφορετικά μοντέλα που αναζητούμε, οι εναλλακτικέ. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό συμβαίνουν αυτά, είναι υπαρκτά και συσχυρίζονται κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναζήτηση εναλλακτικών. Αλλά σε πολλά δεν υπάρχουν εναλλακτικέ από τα πειράματα σε ζώντα ζώα. Αυτό καθίσταται απολύτω σαφέ. Το πλαίσιο λοιπόν που έχουμε σήμερα είναι καλύτερο ή χειρότερο από ότι στο παρελθόν η απάντηση για μένα είναι απόλυτα σαφή. Και επίση και για του επιστήμονε εδώ πολλέ είναι διαφορέ, το ομολογώ. Ακούσαμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, αλλά αναφερθήκαν και οι ομοιότητες. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι χρησιμοποιείται, πότε, με ποιο τρόπο, για να έχουμε τη σωστή επιστημονική προσέγγιση. Ευχαριστώ και... Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι στη δεκαετία του 80 στο Κοινοβούλιο της Δανίας όταν ήμουν βουλευτής για πολλά χρόνια είχαμε φτιάξει έναν πολύ πιο αυστηρό νόμο από ότι η οδηγία αυτή. Ήταν, απαγορευόταν να επιβάλλει κανείς πόνο στα ζώα και έπρεπε να χρησιμοποιούν αναλυτικά κτλ. Αυτό ε, πολλές φορές ε, οδηγεί στην χρήση περισσότερων τύπων ζώων, περισσότερων ειδών. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια απόλυτα ικανοποιητική λύση. Πάντως ε, η πρόταση αυτή την οποία είχαμε κάνει ήταν πολύ πιο αυστηρή από την ισχύουσα οδηγία. Διαρωτώ λοιπόν, Τώρα που διαβάζω τη συγκεκριμένη οδηγία, βλέπω ότι υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις απαιτείται περισσότερος χρόνος συζήτησης, αλλά γιατί να μην υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία όπως αυτή που είχαμε τότε στη Δανία. Ήταν πραγματικά αυστηρή η νόμη και είχαμε αρνηθεί πολλές ε, μορφές έρευνας με ζώα. Προσπαθήσαμε λοιπόν εμείς να μην σταθούμε στα θέματα κριτικής, ζητήσαμε να υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια η οποία είναι απαραίτητη και στα πλαίσια των ε, κλινικών δοκιμών για ανθρώπους το επιβάλαμε και στην αντίστοιχη νομοθεσία για τα ζώα τότε. Σας ευχαριστώ και από την Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα να ζητήσω από την εμπειρογνώμονα που έχετε δίπλα σας λέγοντας ότι το πρώτο ζώο πάνω στο οποίο ε, ε έγιναν δοκιμές ήταν ο άνθρωπος γιατί το 92% των φαρμάκων που περνούν από τα ζώα δεν περνούν στους ανθρώπους, δεν, είναι, ε, δεν επιβεβαιώνονται από τη χρήση στους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικά εδώ μπροστά μας ε, την ε, το απειλητικό φάσμα ε, της φάρμας των ζώων. Εδώ έχουν αρχίσει να βλέπουμε ότι τα ζώα αποκτούν υπερφυσικές δυνάμεις. Και φοβάμαι ότι και οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν την απαιτούμενη διαφάνεια Λοιπόν και η ίδια η ΕΦΣΑ ε, ε, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και ο Όμπουτσμαν της έχει ζητήσει της υπηρεσίας για τα τρόφιμα να είναι πολύ πιο ε, διαφανής και να μην υπάρχουν επικαλύψεις συμφερόντων. Και δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε το λεγόμενο business της ασθένειας όπου και τα νοσοκομεία προσπαθούν να κερδίσουν με παράνομο τρόπο. Κοιτάξτε σας παρακαλώ πολύ ο επόμενος. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που υποστήριξαν την πρωτοβουλία και τους εμπειρογνώμονες που ε, από αυτά που λένε συμπεραίνουν ότι μπορούμε να θέσουμε τέρμα στις, ε, στα πειράματα σε ζώα. Επιτρέπεται πλέον ε, να υπάρχουν δι, δυνατές και ικανοποιητικές εναλλακτικέ μέθοδοι, η τοξικοδυναμική παραδείγματη μέθοδος, ε, μέθοδοι καινοτόμοι, μέθοδοι αποτελεσματικές που μπορούν να δημιουργήσουν και θέσει εργασία και ταυτόχρονα μα επιτρέψουν να θέσουμε τέρμα στα δυνατών ζώων. Η κυρία Γκροστέτα ανησυχεί για τα κέντρα ερεύνη και τα προϊόντα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Θα πρέπει να γίνεται η σωστή επισήμανση των προϊόντων για να μην κινδυνεύουμε να φύγουν τα ερευνητικά κέντρα από την Ευρώπη για να πάνε να κάνουν τα πειράματά του αλλού. Μπορούμε απλώ εδώ να λέμε ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική επισήμανση. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως κάθε πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, στο πνεύμα και το άρθρο 13 της συνθήκης, είναι πολύτιμη. Και πιστεύω ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι αφού υπάρχει οδηγία και εφαρμόζεται πρέπει οι διατάξει τη να υλοποιούνται. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι δηλαδή δεν τηρούνται οι όροι της ε, νομοθεσίας. Ίσως χρειάζεται να υπάρξει κάποιος έλεγχος από εθνική ή και ευρωπαϊκούς φορείς στην τήρηση των όρων της. Εμείς στην Πολωνία, παραδείγματι, επεξεργαζόμαστε νέο νομοθέτημα για τα πείραματα στα ζώα. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι στις επιτροπές δεοντολογίας επικρατούν και τις καθοδηγούν εκείνοι που έχουν συμφέρον από τα πειράματα στα ζώα. Πρέπει λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή να γίνεται η επαλήθευση του σεβασμού. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Την κυρία Μπαρέση Μουσή να πάρει το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω διάφορα σημεία που προκύπτουν από τη συζήτηση. πρέπει να κοιτάξουμε την πρόοδο της εναλλακτικής μεθόδους Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τις ε, μεθόδους και τη τεχνολογία. Θα επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα. Ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε περισσότερη έρευνα στις εναλλακτικέ και για να απαντήσω σε μια από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Το ορίζον 2020 είναι βεβαία πως μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή υποβολής αιτήσεως για υποστήριξη έρευνας σε εναλλακτικέ μεθόδους ή μεθόδους βελτίωσης των μοντέλων με ζώα. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτό που υπόθηκε νωρίτερα για τον ιό του AIDS, HIV που τον γνωρίζω εδώ και χρόνια. Είπατε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο. Ναι, συμφωνώ πολύ Αλλά πιστεύετε πράγματι ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από τα πρότυπα ζώων και νομίζω ότι αυτή η προόδος στην έρευνα για τον ιό του AIDS δεν έχει καμία σχέση των αντίων. Επειδή έχουμε όλα αυτά τα χρόνια συλλέξει αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε λοιπόν να βρούμε αντισώματα που είναι αποτελεσματικά στα ζωικά μοντέλα και από τις τελευταίες επιστημονικές καταγραφές επιβεβαιώνουν απολύτως τα δεδομένα από ζωικά μοντέλα και μάλιστα μαϊμούδες. Αυτά για την κυρία Σάντερ. Αν σήμερα μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα από την έρευνα, και εναλλακτικά πρότυπα. εάν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αποτελέσματα για εμβόλιο και θεραπεία, γιατί ο, ο ασθενής σήμερα περιμένει μια απάντηση για θεραπεία, εγώ δυστυχώς σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσω ότι σήμερα δεν είναι δυνατόν. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταφέρουμε, αλλά σήμερα όχι. Μια άλλη ερώτηση για το αν μεταφέρονται τα δεδομένα από ζωικά μοντέλα στον άνθρωπο. Ναι, σας ανέφερα νωρίτερα. Μάλλον εσείς αναφέρατε τον ε, ιό έμπολα. Τρεις θεραπείες που δοκιμάστηκαν πρόσφατα για τον έμπολα έχουν επιβεβαιωθεί στον άνθρωπο. Μια από αυτές είναι ένα κοκτέιλ αντισωμάτων που σε μακάκο αποδεικνύει 43% αποτελεσματικότητας. Σε μοντέλο μακάκου με δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από δοκιμές σε άνθρωπο, 45% ήταν η επιτυχία, η αποτελεσματικότητα μάλλον, του κοκτέιλ αυτού. Άρα ναι, μπορεί να γίνει μεταφορά, εάν χρησιμοποιείται σωστά το μοντέλο. Στις βέλτιστες συνθήκες με βάση το βέλτιστο σχεδιασμό και αυτό έχει κρίσιμη σημασία. Εν τέλει θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να αντιτασσόμεθα σε εναλλακτικέ μεθόδους, ζωικά μοντέλα, κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Χρειαζόμαστε και τις τρεις επιλογές. Είναι αλληλοσυμπληρούμενες σήμερα και πιστεύω ειλικρινά, ελπίζω ειλικρινά όπως όλοι σας, ότι κάποια μέρα θα έχουμε καλύτερες μεθόδους, καλύτερες προσεγγίσεις για να μειώσουμε ακόμη και να αποκλείσουμε, να σταματήσουμε όλος διόλου κάποιες δοκιμές και να μπορούμε να προβλέπουμε τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους με τρόπους. Και πάλι απευθύνω έκκληση σήμερα με κίνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Horizon 2020 είναι η καλύτερη λύση. Μιλάμε για την καινοτομία. Ε, χρειαζόμαστε την καινοτομία σε επαρκή βαθμό για το μέλλον. Χρειαζόμαστε την καινοτομία για να έχουμε καλύτερα μοντέλα ζωικά. Με ανησυχεί όμω το ότι στην προκήρυξη του ορίζον 2020 δεν υπάρχει αναφορά σε λοιμώδεις νόσους. Όταν αναδεικνύονται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο λοιμώδεις νόσοι όπως αυτή του ιού έμπολα. Απευθύνω λοιπόν και εγώ έκκληση. Πρέπει να καταστήσουμε σαφέ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η προκήρυξη η ευρωπαϊκή θα είναι τέτοια ώστε να ανταπακρίνεται στην ανάγκη για τη βελτίωση της υγείας τους των ζώων και των ανθρώπων. Są pytania do pana, do pana dyrektora Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αντιδράσω σε κάποιες από τις προτάσεις που άκουσα στη συζήτηση που προηγήθηκε γύρω από την οδηγία. Άκουσα ότι η οδηγία δεν επιτρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες. Αν διαβάσετε το άρθρο 2 θα καταλάβετε ότι επιτρέπεται η λήψη αυστηρότερων μέτρων ιδιαίτερα για τις χώρες που είχαν τα μέτρα αυτά. Αυτό χρησιμοποιείται από διάφορες χώρες οι οποίες ενημέρωσαν ότι θα διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα. Η νομοθεσία η Δανέζικη σχετικά με τη χρήση ανεμφυσίας. Ε, θα ήθελα να δείτε το άρθρο 14 της οδηγίας είναι κάτι που και αυτό ανήκει στην οδηγία του 2010. Και τέλος άκουσα ότι θα ήταν αδύνατο για τους επιστήμονες να αμφισβητήσουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από επιστημονικά ευρωπαϊκά όργανα. Η οδηγία αυτή όπως και όλες οι άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να αμφισβητηθούν από οποιοδήποτε πολίτη. Μπορεί κανείς να προσφύγει απευθείας στα δικαστήρια, μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να περάσει από την Επιτροπή Αναφορών. Υπάρχουν τρόποι και οδοί όπως και για όλες τις άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις αμφισβήτησης. Έχει σημασία λοιπόν να συνεργαστούμε στα πλαίσια της σωστής εφαρμογής τους, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους η συγκεκριμένη οδηγία έχει θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα από πλευρά των οργανωτών θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ρέης. Ευχαριστώ πολύ. θα ήθελα πράγματι να δώσω κάποια επιστημονικά στοιχεία για να μπορέσετε να κρίνετε καλύτερα αυτά τα οποία είπε και η κυρία Σύνωση και την ευχαριστώ για την παρουσίασή της η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αλλά δεν με έπεισε. Είδα τις δημοσιεύσεις της κυρίας Σύνωση, είναι 270 και πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις έχουν σχέση με τα προβλήματα μεταφοράς του ιού του AIDS από τη μητέρα στο παιδί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και τη συγχαίρω για τις προτάσεις της σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Γενικότερα, αν μπορούσαμε να θεραπεύσουμε το AIDS, δεν θα μας ανησυχούσε η μεταφορά του ιού ανάμεσα στο μητέρα και στο παιδί. Γιατί λοιπόν να μην αναπτύξουμε μια θεραπεία κατά του AIDS. Η κυρία Σινουσή εδώ και 30 χρόνια κάνει έρευνα για να βρει ακριβώς αυτά τα φάρμακα. Έχουν υπάρξει δεκάδες χιλιάδες μελέτες ταυτόχρονα στον υπόλοιπο κόσμο και προς το παρόν δεν έχουμε βρει λύση. Πρέπει να τεθεί λοιπόν το θέμα αυτό. Όταν ήμουν υπεύθυνο των εργαστηρίων Παγιάς, είχαμε αναπτύξει κάποιες μεθόδους και όταν είδαμε ότι μετά από τρεις-τέσσερις ε, ε, αποτυχίες ε, αλλάζαμε το πεδίο παρέμβασης. Η κυρία Συνουσή όμως χρησιμοποιεί την ίδια υπόθεση. Μελετά στους μακάκους και στους χιμπατζίδες επίσης τον ιό όχι του HIV αλλά του SIV που είναι το AIDS του πυθίκου. Ε, δεν είναι όμως το ίδιο οι δύο αυτές ασθένειες. Και τα αποτελέσματά σας αποδεικνύουν αδιαφυσβήτητα και χωρίς να το ξέρετε ότι το HIV και το SIV δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να κάνω μια υπόθεση λογική για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα. Να προσπαθήσει κανείς να φτιάξει ένα εμβόλιο για το AIDS είναι αδύνατον. Έχετε ένα στόχο που μετακινείται συνεχώς και με μεγάλη ταχύτητα γιατί μεταλλάσσετε μονίμως. Όταν εσείς φτιάξετε ε, το εμβόλιο για ένα δεδομένο ιό, ο ιός θα έχει ήδη αλλάξει. Αντίθετα, όταν βλέπετε από κοντά τους μηχανισμούς που επιτρέψουν σε αυτό τον, ε, τον ιό να αποφύγει ε, το σύστημα αυτό, τότε ε, θα έχετε κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας έχει καταθέσει ένα δίπλωμα έβρεση τεχνίας για μια θεραπευτική αντιμετώπιση του AIDS που επιτρέπει να φεύγει ο ιός από το σώμα του ασθενούς. Το δίπλωμα αυτό προτάθηκε και στην φαρμακευτική βιομηχανία, της οποίας υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ, και μας είπανε κάντε τις κλινικές δοκιμές, ε, ολοκληρώστε ε, πριν έλθετε σε μας. Το ΣΕΝΕΡΕΣ ε, δεν έχει τις αρμοδιότητες να κάνει τέτοιου είδους τεχνικές μελέτες. Εγώ ήρθα σε επαφή με τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες και όλες μου απάντησαν το ίδιο πράγμα μας είπαν ότι το AIDS για μας είναι ένα business που αντιπροσωπεύει 36 δις κατέτος και δεν έχουμε καμία διάθεση να σταματήσουμε την τροφοδοσία την οικονομική αυτών των επιχειρήσεων. Κυρία Σίνουση μπορείτε να το σχολιάσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Ε, με τα χαράς να το σχολιάσω. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν εκπροσωπώ καμία φαρμακοβιομηχανία. Γιατί εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω εργαστεί για φαρμακοβιομηχανία. Είμαι επιστήμων. Εργάζομαι για το πανεπιστήμιο. Δεν έχω χρηματοδοτηθεί ποτέ από τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω. Δεύτερον, νομίζω ότι δεν έχετε μελετήσει πολύ προσεκτικά τη βιβλιογραφία μου. Εδώ και 33 χρόνια έχω εργαστεί. Δεν με απασχολεί το θέμα της μετάδοσης ε, του HIV ούτε η έρευνα για τα εμβόλια. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει θεραπεία για τον ιό του AIDS. Και ξέρετε, δεν θεωρείται πλέον μοιραία θανατηφόρα νόσος το AIDS. Μπορεί να ζήσει ένας ε, ασθενής με AIDS. Πάνω από 4 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο έχουμε αποφύγει χάρη σε αυτή τη θεραπεία σήμερα είναι μια χρόνια λίμωξη που θεραπεύεται το AIDS και με τη θεραπεία αυτή και οι θάνατοι του ασθενούς, των ασθενών αποφεύγονται. Το δε προσδόκιμο ζωής είναι πολύ παρόμοιο με το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων που δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Όμως η θεραπεία αυτή είναι και πρόληψη, γιατί μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο έμβριο. Και χαίρομαι πολύ που δεν έχουμε χώρες όπου η πρόσβαση θεραπεία δεν είναι διαθέσιμη. Και πια δεν μεταδίδεται ο ιός ε, ένα ε, το από τη μητέρα στο παιδί. Όμως, σίγουρα, από την άλλη πλευρά, πολύ δύσκολα μπορεί να διατεθεί σε όλους αυτή η θεραπεία. Έχουμε μόνο ένα 40% στον κόσμο προθετικών που έχουν πρόσβαση στον, σε αυτή τη θεραπεία, το 60% δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι μένει πολύ πρόοδο να γίνει και σήμερα αυτή είναι η δουλειά μου. Προσπαθώ να καταλάβω το μηχανισμό με τον οποίο ορισμένοι, ορισμένοι ασθενείς ελέγχουν με φυσικό τρόπο την λίμωξη αυτή. Και αυτό τελείως διαφορετικό από αυτό που εσείς είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαγεσινουσή. Ολοκληρώνεται έτσι και ο δεύτερος γύρος της συζήτησης. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και την καθηγήτρια Μπαγεσινουσή και έρχομαι στο τρίτο γύρο. Η κυρία Μακάιβορ είναι η ομιλήτρια από τη Human Society International να έρθει παρακαλώ στο βήμα μέχρι να έρθει στο ε, βήμα να μιλήσω για ένα πρόγραμμα ελκυστικότητας της Ευρώπης σε σχέση με την ε, βασική έρευνα. Ίσως η Ήπειρος αυτή καταστεί καθόλου ελκυστική τελικά για τους επιστήμονες. Οι δοκιμές, η έρευνα ε, γίνονται αλλού, όπου επικρατούν λιγότερο περιοριστικοί νομικοί όροι. και οι επιλογές είναι πολύ δύσκολες σίγουρα. Δέκα λεπτά έχετε κύριε Μακάβρο στη διάθεσή σας. Καλό απόγευμα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να συγχαρώ του διοργανωτέ τη πρωτοβουλία των πολιτών που συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφέ για να σταματήσουν τα πειράματα κατά των ζώων. Θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο σε δράσεις και όχι τόσο σε επιχειρήματα που έχουμε ακούσει. Γιατί υπάρχουν δράσεις που μπορούν να, να αναλυθούν αμέσως, ενώ κάποιες μπορούν να μείνουν για το μέλλον. Πέραν των δράσεων που μπορεί να έχουν να εκφράζουμε κάποιες προσδοκίες, υπάρχουν δράσεις που απορρέουν από υποχρεώσεις, ενισχύ και μπορούν αυτές να μειώσουν και να περιορίσουν τα πειράματα στα ζώα, ήδη τώρα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Γίνανε πολλές συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πειράματα στα ζώα. Τι προξένουν στα ζώα και πώς μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Αν γυρίσουμε όμως πίσω στο 1993 όπου ανέλαβαν δράση οι πολίτες για να σταματήσουν τα πειράματα εις βάρος των ζώων για καλλιτικά. Είναι σαφές ότι ο πόνος που υφιστούν τα ζώα δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από την ανάγκη παραγωγής καλλιτικών. Είδαμε λοιπόν μετά τις πιέσεις των πολιτών την ανάληψη δράση και από τις κυβερνήσεις και την απαγόρευση των πειραμάτων σε καλλιτικά, ε, για καλλιτικά και τη πώληση των προϊόντων αυτών. Είδαμε λοιπόν ότι άλλαξαν πολλά πράγματα, αλλά ίσως υπέφερε η επιλογή του κανονιστικού θα πω ε, συστήματος ε, δοκιμών το regulatory testing συγκεκριμένα. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν των πολιτών έχει μεταφέρει την εστίαση της προσοχής σε όλα τα είδη πειραμάτων σε ζώα και τη βιοιατρική έρευνα συγκεκριμένα. Αλλά ας κοιτάξουμε το regulatory testing και το λόγο για τον οποίο οι πολίτες, οι, οι πολιτικοί έχουν τόσο πολύ προσέξει την υπόθεση. Με την πρόταση του 2001 με το REACH Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μέχρι και 5 εκατομμύρια ζώα μπορούσαν να πέφτουν θύματα πειραμάτων. Έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια. Και εγώ προσπαθώ να εξασφαλίσω την τήρηση των υποχρεώσεων. Όπου υπάρχουν δηλαδή, τουλάχιστον όπου υπάρχουν ελλακτικέ, να μην γίνονται πειράματα σε ζώα. Αυτό είναι το πιο απλό. Να αντικαθίστανται τα πειράματα σε ζώντα ζώα από άλλε εξίσου καλέ μεθόδου. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε, τι κάνουμε στα υπόλοιπα. Θα μπορούσα να μιλήσω και άλλο για το Ρίτσο, αλλά δεν έχω χρόνο. Και προχωρώ. Τα τελευταία 15 χρόνια είδαμε την εμφάνιση αυτής της νέας οδηγίας, της υπερθυμών 63, η οποία λέει ότι μπορεί να βελτιώνεται η εφαρμογή και οι όροι από τους οποίους εφαρμόζονται τα πειράματα. Ταυτόχρονα όμως λέει ότι εξασφαλίζονται και δημιουργούνται διάφοροι τρόποι να προαχθεί η επιστήμη. Ας ξαναγυρίσω όμως την βιοιατρική έρευνα. Η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να επανέλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η βιοιατρική έρευνα και να μιλήσουμε για τα εκατομμύρια αυτών ζώων που χρησιμοποιούνται για βιοιατρική έρευνα στην Ευρώπη, σε πειράματα. Είναι η στιγμή της καμπής, το σημείο καμπής. Είναι η πρώτη φορά που συζητείται με αυτού τους όρους και στο Κοινοβούλιο η χρήση ζώων σε πειράματα για τη βιοιατρική έρευνα. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη κρίση. Σας έχω αυτό το έντυπο στην είσοδο που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποτύχει οι έρευνες στην ιδιοιατρική που χρησιμοποιούν σώα στο στόχο της βελτίωσης της υγείας των ανθρώπων. Εξετάζουμε δηλαδή τι σημαίνει ζωικό πρότυπο, ζωικό μοντέλο για με ανθρώπινη νόσο, που μπορεί να μην εμφανίζεται με φυσιολογικούς όρους στα ζώα, άρα πρέπει να προξενηθούν σύμπτωμα στα ζώα, συμπτώματα στα ζώα, για τα οποία συμπτώματα αναζητώνται μετά θεραπείες. Και μετά θα γίνουν τα τοξικολογικά τεστ. Μετά λοιπόν από αυτές τις δοκιμές και τις τοξικολογικές αποδεικνύεται ότι 95% των φαρμάκων αποτυγχάνουν την κλινική δοκιμή στον άνθρωπο. Η τοξικολογία και η αποτελεσματικότητα είναι μη αξιόπιστες δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για την αποτελεσματικότητα, αλλά περισσότερο για το μέχρι τώρα. Ας κοιτάξουμε τώρα και την αποτελεσματικότητα. Στη σκλήρινση κατά πλάκα 49% των φαρμάκων έχουν αποτύχει στις κλινικές δοκιμές. Στο άσθμα, ύστερα από δεκαετίες πειραμάτων στα ζώα, έχουμε μόνο δύο νέες κλάσεις φαρμάκων. Έχω πολύ μακρό σκελή κατάλογο να παρουσιάσω. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τι εργαλεία έχουμε στη θέση μας ένα από αυτά το προσφέρει συνθήκη. Το άρθρο 13 μας υπενθυμίζει ότι η ευζοία των ζώων είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άρθρο 8 της Οδηγίας 2010, κάθετος 63, μας υπενθυμίζει ότι η ευζοία των ζώων είναι αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αρχή που δεν μπορούμε να λησμονούμε, δεν μπορούμε να αγνοούμε μια αρχή που πρέπει να μας κεντρήσει όλους για να λάβουμε δράση. Πώς μπορούμε λοιπόν τις αξίες αυτές να τις ε, θέσουμε, να τις μεταστράψουμε σε δράση. Έχω ετοιμάσει μια διαφάνεια για ένα πολύ απλό πράγμα. Από τα 11,5% ε, εκατομμύρια ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2% υφίσταται βαρέα λεγόμενα πειράματα. Σας δείχνω εδώ τις, ε, τα ηλεκτροσόκ, την απομόνωση για παρατεταμένες περιόδους, την ε, ακινητοποίηση προκειμένου να προξενηθούν ε, έλκη, κοιλιακά ή καρδιακή ανεπάρκεια, υποχρεωτική κολύμβηση ή ασκήσεις εξάντλησης. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, μα πώς το μετράτε αυτό, τι σημαίνει πόνος, εξάντληση κτλ. Ναι, υπάρχει τρόπος μέτρησης και μπορούμε να προχωρήσουμε. Η οδηγία ίδια λέει ότι τελικός στόχος είναι η πλήρης αντικατάσταση των διαδικασιών των ζώων. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν ώστε να αντικατασταθούν πλήρως οι διαδικασίες των ζώων. Μπορούμε να βρούμε νέες λύσεις. Υπάρχει ένα, ένα βρετανικό επραδείγματι σχέδιο που έχει προτείνει και με τη ρυθμιστική αρχή για τα πειράματα στα ζώα και με σώματα υπεύθυνα για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, ε, υγειονομική των τροφίμων κτλ. Λύσεις και συνενέσεις. που μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικέ και ευζοία. Γιατί το 95% της αποτυχίας είναι καταδικαστικό για τις εταιρείες τις φαρμακευτικές όπως και για τα πειράματα. Κίνητρα λοιπόν, αξιολόγηση, αναδρομική αξιολόγηση και έλεγχος αν επαληθεύθηκαν οι στόχοι του πειράματος. Η Επιτροπή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αυτοί είμαστε εμείς πρέπει να τα κοιτάξει όλα αυτά στην αναθεώρηση της οδηγίας για να δει τι έχει επιφέρει και αν υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς με στόχο και αρμοδιότητα να καλύπτει τις εναλλακτικέ και στη βιοιατρική, απεκτάθηκε το πεδίο δράσης του 2010, αλλά πάνω απ' όλα την αντικατάσταση των πειραμάτων στα ζωά. Και επίσης το Βρετανικό αυτό σχέδιο υποδεικνύει πως μπορεί να υπάρχει ένας εντηρητισμός σε επίπεδο επιστημόνων, ελεγκτών ή αναθεωρητών των συστημάτων. Ένας εντηρητισμός τον οποίο πρέπει να ανατρέψουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα εκ μέρους των εφών πολιτικών ομάδων. Καταρχάς ο κ. με τρία λεπτά στη διάθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον και κοινωνικό ενδιαφέρον. Και να ευχαριστήσω την κυρία Μακάιβορ για την πληρότητα της παρέμβασής της. Για αυτά τα θέματα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε βάθος η οποία συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι προκατελημένη. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στον επιστημονικό κόσμο που δείχνουν ότι είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια πραγματική λύση. Όταν ένα εκατομμύριο πολίτες προτείνουν μια τέτοια αναφορά, το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους ακούσει και να λάβει υπόψη την πρότασή Δεν είναι εύκολο να συλλέξει κανείς ένα εκατομμύριο υπογραφών. Συγχαίρω λοιπόν τους οργανωτές για την προσπάθειά τους και η επιτυχία τους είναι μια νίκη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αποδεικνύει η πρωτοβουλία ότι οι πολίτες έχουν ε, τα μέσα να καθορίζουν την κοινοτική πολιτική και πολύ συχνά οι πολίτες, ο συνήθως μάλλον οι πολίτες είναι ένα βήμα μπροστά από τους πολιτικούς. Ζητούν να υπάρξει πάυση ισχύω της συγκεκριμένη οδηγίας, να παρουσιαστεί μια νέα πρόταση η οποία να απαγορεύει τα πειράματα σε ζώα. Είναι ένα θέμα αυτό εξαιρετικά σημαντικό και για λόγους δεοντολογικούς και λόγω της διτής χρήσης αυτών των πειραμάτων, κάτι που υπογράμμισαν οι προλαλήσαντες. Ζητάμε λοιπόν από τα κοινοτικά όργανα να πάρουν μέτρα προστατεύοντας την υγεία των ζώων. Νομίζω ότι η διαφάνεια την οποία είδαμε πριν είναι εξαιρετική. Η υγεία των ζώων πάντα ήταν μια προτεραιότητα. Το λέγει άλλωστε και το 12 της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε δύο θα έλεγα τομείς. Πρώτον, να ελέγξουμε σωστά την χρήση των ζώων μέσω πρόθεσμα και ε, να αναζητήσουμε εναλλακτικέ λύσεις όπως ακριβώς είπε η κυρία Μακάιβαρ. Και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πληροφορίες ε, για τις χρήσεις των συγκεκριμένων μεθόδων με ε, ζώντα ζώα και να είναι σε θέση οι πολίτες να γνωρίζουν το τι συμβαίνει στα διάφορα εργαστήρια τα οποία κάνουν τα πειράματα. Θα πρέπει επίσης σε μια δεύτερη φάση να προωθήσουμε τις εναλλακτικές μεθόδους. Έχω τέσσερα λεπτά και κλείνω όπου να είναι, λέει ο κύριος Καπούτο. Θα πρέπει οι νέες μέθοδοι να προτιμούνται εφόσον είναι διαθέσιμοι. Θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές και οι ερευνητές δεν θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποφασίζουν ε, την επιλογή. Ε, τα εναλλακτικά ε, προ στιγμήν δεν θα είναι βέβαια ε, τα εναλλακτικά συστήματα τα μοναδικά σε μια πρώτη φάση. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πρώτο καλό βήμα να προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε. Τώρα προσπαθώντας να αντικαταστήσουμε την, αποφάσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από νομικές αποφάσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα σε πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ κύριε καστάλτη. Ο κύριος Καστάλτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις στη συγκεκριμένη οδηγία. Προβλέπεται μια διοικητική απλοποιημένη διαδικασία μέσα από την οποία τα κρατη μπορούν να δώσουν άδειε έρευνα ισχύω 5 ετών. Ε, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες επεξηγήσεις και προϋποθέσεις, άρθρα 40 και 41 της συνθήκης, με συγκεκριμένες μεθόδους έρευνας αλλά δυστυχώς ε, δεν ζητείται να υπάρξει μια μη τεχνική ε, παρουσίαση του προγράμματος. Κανονικά θα έπρεπε με ανώνυμο τρόπο να δώσουν μια σειρά πληροφοριών που είναι για μας σημαντικές για τους στόχους του προγράμματος και για τον αριθμό των ζώων και τα είδη των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν και αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια στα κράτη-μέλη. Τίθεται λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα διαφάνειας γιατί δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει στα εργαστήρια και τα σκάνδαλα βίας εις βάρος των ζώων είναι πάρα πολύ συχνά δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς μπορούμε λοιπόν να επανορθώσουμε την κατάσταση αυτή ε, εφόσον ε, γνωρίζουμε ότι οι επίσημες στατιστικές για την απλοποιημένη διαδικασία και τη χρήση της διαδικασίας αυτής ε, γίνεται με στρεβλό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να ξεπεραστεί η οδηγία αυτή, πρέπει να έχουμε σαν βασικό στόχο το να ακούσουμε τη φωνή του Ευρωπαίου πολίτη, δεν είναι μια επιλογή. Είμαστε υποχρεωμένοι για ένα εκατομμύριο καλούς λόγους. Ευχαριστώ. Μάκερ. Eh, Ευχαριστώ την κυρία Μακάιβορ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θέλω επίσης με την ευκαιρία να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να πω ότι θέλω να προσεγγίσω το θέμα με ανοιχτό πνεύμα. Μου αρέσουν και οι άνθρωποι και τα ζώα. Εγώ λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να απαγορευτούν εντελώς οι δοκιμές σε ζώα, αλλά να μειωθούν στο δυνατόν περισσότερο και ίσως ενδεχομένως κάποιοι να καταργηθούν. Ένα ερώτημα έχω. Η συμφωνία TTIP, τι, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ενδεχομένω. Είπατε ότι η καλή μεταχείριση των ζώων είναι μια από τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία TTIP θα επηρεάσει μάλλον σημαντικά ε, τα ζώα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για επιστημονικές δοκιμές. Και Ίσως υπάρχουν θετικές επιπτώσεις. Η TTIP, Διατλαντική Συμφωνία Μπορεί και Επενδύσεων, έχει να κάνει με εναρμόνιση προτύπων και κανόνων για εμπορικούς σκοπούς υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Όμως, τίθεται και το θέμα της αποφυγής αλληλεπικάλυψης και εφαρμογή διαφορετικών προτύπων. Θα μπορούσε δηλαδή η συμφωνία TTIP να συμβάλλει στην εφαρμογή της αρχής των τριών R, άρα να οδηγήσει σε μείωση των ε, δοκιμών σε ζώα. Ποια είναι η άποψή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Εύη. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ ότι καλύτερο σε αυτή την πρωτοβουλία κατά των πειραμάτων με ζώα και να υπάρξει μια συγκεκριμένη απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι αντίστοιχη με την αντίστοιχη πρωτοβουλία για τα νερά, για τα ύδατα, ε, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία αυτή με τον σωστό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την εκ νέου χρήση των ζώων σε πολλαπλά πειράματα. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα όριο στις ελαφρές ή μέτριες διαδικασίες τις οποίες υφίστανται τα ζώα. Οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες και περιλαμβάνονται και στην προσθήκη 8, στο παράρτημα συγγνώμη 8 ε, της οδηγίας. Προβλέπει η οδηγία ότι η σοβαρότητα καθορίζεται από το επίπεδο πόνου, άγχους και αγωνίας την οποία αισθάνεται το ζώο. Η οδηγία επιτρέπει για πρώτη φορά αντίθετα με την οδηγία του 86 και εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί δηλαδή παναχωρήσαμε αντί να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός με μια νέα οδηγία ότι επιτρέπονται λοιπόν και άγρια να γίνονται τέτοιου είδους ε, πειράματα και σε σε αδέσποτα ζώα, σκύλου και γάτες. Λοιπόν, θα πρέπει πράγματι η οδηγία να προστατεύει την ευημερία των ζώων και όχι το αντίθετο. Ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ζώα νιώθουν τον πόνο. Γι' αυτό τα 11,5 αυτά εκατομμύρια ζώα που είναι στα πειράματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαράδεκτα. 0,5 μόλις λιγότερα ζώα χρησιμοποιούνται σε πειράματα από τα τελευταία 5 χρόνια, 7 χρόνια. Αυτό δεν είναι πρόοδος και γι' αυτό ιδιαίτερα χαίρομαι για την πρωτοβουλία των πολιτών γιατί χρειάζεται πολιτική πίεση για να συνεχίσουμε. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο εσείς προτείνατε, αναφέρατε για το πού γίνονται τα πειράματα έχει πολύ μεγάλη σημασία. 90% στη βιοιατρική ή αντίστοιχα και μόλις 10 και λιγότερο της 100 στα ρυθμιστικά, στις ρυθμιστικές δοκιμές, regulatory testing. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι με καταπλήσουν αρνητικά ορισμένοι συνάδελφοι και ο κύριος Ταραμπέλα ιδιαιτέρως το να βάζουμε να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις για τα πείραματα των ζώων είναι απαράδεκτο κυρίως να λέμε ότι άμα τα απαγορεύσουμε καταδικάζουμε τόσους ανθρώπους σε θάνατο. Και ώστε οφείλει συγγνώμη, νομίζω, για τα λόγια αυτά. Η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρει πολύ στα σοβαρά την πρωτοβουλία αυτή και αναμένω από την Επιτροπή και είμαστε πολλοί όπως εγώ που περιμένουμε συγκεκριμένε απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία 2010-63 δεν ξέρω αν θα πρέπει πράγματι αμέσω να καταργηθεί. Αλλά είναι βέβαιο πω η οδηγία αυτή χρειάζεται βελτίωση. Και το δεύτερο, να, κάνουμε, να συνεχίσουμε ε, περισσότερα χρήματα στην εναλλακτική έρευνα. Έχουμε όμω πολλά προβλήματα ακόμη. Ότι δεν τηρείται σωστά η οδηγία για τα καλλιντικά. Και αν είναι γνωστές Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κάποιοι άλλοι έχουν ξεπεράσει τον χρόνο του Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου. Άλλοι λοιπόν. Ξέρουμε λοιπόν ότι στην οδηγία για τα καλλιτικά υπάρχουν παραθυράκια τα οποία αξιοποιούνται ακόμη και θέλω να την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς είναι δυνατόν να δέσουμε ένα τέρμα σε αυτήν την κατάσταση γιατί δεν είναι αποδεκτή. Έγινε λόγος επίσης για συντηρητισμό. Μιλήσατε για συντηρητισμό των επιστημόνων και των ερευνητών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πατάξουμε το συντηρητισμό Ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιοι εκπρόσωποι τροπών που του έδωσα το λόγο για περισσότερη ώρα να δώσω τώρα στον κύριο Τσούλο το λόγο. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά επιχειρήματα στα τελευταία δύο πάνελ. Η προηγούμενη ομιλήτρια είπε ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρώπη να ενισχύσει την έρευνα της αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων. Τώρα ακούσαμε ότι οι υπάρχοντες κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί. Νομίζω ότι έχουμε δύο δυνατότητες επίσημα μπροστά μας, δύο δρόμους να ακολουθήσουμε. Πρώτον, αυτό όμως που μπορούμε πράγματι να υποστηρίξουμε είναι η φωνή των πολιτών, τίποτα άλλο, δεν υπάρχει αναλλακτική λύση. Ελείπει η πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο η οποία θα πρέπει και οικονομικά να υποστηρίξει και σε επίπεδο διακανονιστικό τη συγκεκριμένη επιλογή των εναλλακτικών μεθόδων. Εμείς είδαμε στα πλαίσια της συνθήκης στο άρθρο 13 ποια είναι η σημασία, υπογραμμίζουμε τη σημασία της ευημερία των ζώων. Αυτές τις ημέρες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται τον κανονισμό για τις ζωονόσους που μεταδίδονται στους ανθρώπους. Στον κανονισμό αυτό έχουν ε, εισαχθεί νέες έννοιες σε σχέση με την ευημερία των ζώων, αλλά σε ελάχιστο βαθμό. Γιατί θεωρήθηκαν ε, οι προτάσεις που έγιναν γύρω από αυτό εκτός θέματος. Πότε θα μας ακούσει τους πολίτες, πότε θα υπάρξει μια πραγματική οδηγία για την ευημερία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ οι εμπειρογνώμων μας. Η κυρία Μακάη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά δικαιολόγητες ε, ελλείψεις οδηγίας, οι ασφάλματα σίγουρα είναι πολλές για την οδηγίες. Η αποστευμένη διαδικασία που αναφέρεται είναι μία ε, ανεπάρκεια. Επίσης, ούτε αφορά την αξιολόγηση των έργων, αν απαιτείται διανόμου μία δοκιμή μπορεί να γίνει, αλλά ε, αν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Ε, θα γυρίσω στο συντηρητισμό αργότερα. Να πω προς το παρόν κάτι για τη συμφωνία TTIP. Τα πειράματα σε ζώα αντιπροσωπεύουν ένα ενδιαφέρον ε, θέμα στο πλαίσιο τη TTIP, γιατί στο πλαίσιο των ρυθμιστικών δοκιμών είναι πλεονέκτημα μεγάλων επιχειρήσεων ε, πολυεθνικών να μειώσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τι δοκιμέ εδώ, γιατί αυτό ε, σημαίνει οικονομίε. Γι' αυτό και υπάρχει όθηση να μειωθούν αυτέ οι δοκιμές στο συμφωνία TTIP δεν, ε, προ, δεν καλύπτεται όμως ε, η νομοθεσία για, τα, την προστασία των ζώων. Οι χαρουρέοι και οι ποντικοί δεν προστατεύονται από την νομοθεσία και σε αυτά τα ζώα γίνονται περισσότερες δοκιμές. Συνολικά η συμφωνία TTIP λοιπόν ε, συνιστά απειλή σε αυτό το τομέα. Θα θεωρούσα επίσης ε, επιπροσθέτως ότι έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόοδο με την οδηγία για τα καλλιντικά. Φοβούμαι ότι η απώλεια δημοκρατίας λόγω της συμφωνίας TTIP θα μειώσει και τι δικέ μας δυνατότητες να εισαγάγουμε νομοθεσία αντίστοιχη ε, με βάση τη δημόσια ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμη. και αυτούς του ε, πολύ χαλαρούς νόμους περί επαναχρησιμοποίηση. Να είναι ντροπή το ίδιο ισχύει και με τις λεγόμενες ρήτρες διασφάλισης που επιτρέπουν πειράματα σε ζώα πιο σοβαρά σε σχέση με τον κατάλογο που σας ε, ε, απαριθμίσα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και φοβούμαι ότι ο, για την ευθύνη ε, μόνο η άσκηση πίσω από τον κλάδο αυτή έχει την ευθύνη γιατί δεν θέλουν καμία απαγόρευση και θέλουν να υπάρχει δυνατότητα να υπερβούν ε, τα επιτρεπόμενα από το νόμο, από το δίκαιο. Και αυτό ε, έχει να κάνει και με αυτές τις αδυναμίες της οδηγίας για την προστασία των ζώων. Μέσω των ερητρών διασφάλισης που θεωρητικά ε, προβλέπουν τη χρήση γραφειοκρατίας, ευθοκρατικών μεθόδων. Σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να σταματήσουμε να είμαστε συντηρητικοί. Πρέπει να συνομιλούμε περισσότερο και εμείς η κοινότητα που είμαστε υπέρ προστασία των ζώων θα πρέπει να δώσουμε στην Κομισιόν ένα συνεκτικό μήνυμα για το ε, ποιος είναι ο στόχος και επιθυμής μας ό,τι αφορά τα πειράματα σε ζώα και πώς θα βοηθήσουμε ε, να αρθούν αυτά τα πολύ αρνητικά ποσοστά, 95% αποτυχίας ε, των δοκιμών ε, αποτελεσματικότητας ή σκοπιμότητας. Και καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας την αύξηση της ευημερίας, τη βελτίωση της ευημερίας. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που δίνει αυτή η οδηγία, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και ευθύνη για την πλημελή εφαρμογή έχουν τα κράτη-μέλη για το πώ εφαρμόζουν κάποιες διαδικασίες. Ε, την αξιολόγηση των έργων, για παράδειγμα, αν οι υπεύθυνοι αξιολόγηση ε, θεωρούν ε, το πείραμα μπορεί να μην επιτελέσει το σκοπό του ό,τι αφορά και τη σχέση κόστου ωφέλου, μπορεί να σταματήσει αυτή η δοκιμή. Το ίδιο αν θεωρούν οι αξιολογητέ ότι υπάρχει καλύτερη επιστημονική εναλλακτική, που στην περίπτωση τη βιοιατρική έρευνα μπορεί να είναι μια άλλη τεχνολογία και να μην προχωρήσει συγκεκριμένη. E, Σα ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε τον τρίτο γύρο της συζήτηση, θα παρακαλέσω τον κύριο Μενάς, έναν εκ των ε, διοργανωτών, για πέντε λεπτά να πάρει το λόγο. Η μεγαλύτερη πρόκληση στην πρωτοβουλία αυτή δεν είναι η επιστήμη αλλά η επικοινωνία. Η βασική ιδέα πίσω από το ECI ήταν να ανέβει το επίπεδο της συζήτησης από το θέμα της ευημερίας των ζώων μέχρι το επίπεδο της εγκυρότητας του προτύπου. Και αυτό έγινε κάτι το οποίο περιορίστηκε στο θέμα της επιστήμης. Βασικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να οργανώσει ε, μια διαβούλευση, όχι με 10 λεπτά ο καθένας, αλλά 3, 4, 5 μέρες για να συζητήσουμε την τεκμηρίωση της επιστήμης με εμπειρογνώμονες από τις δύο πλευρές. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια σοβαρή συζήτηση, τότε φοβάμαι ότι ε, ε, περιφρονούμε αυτά τα οποία ζητούν αυτοί οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους. Και επίσης αγνοούμε και αυτούς οι οποίοι θέλουν φάρμακα με προσωπική έγκριση, αποδοχή αν θέλετε. Πάρτε το παράδειγμα του Μποτόξ. Το γνωρίζετε πολύ, λίγοι το χρησιμοποιείτε είναι ίσως το πιο η πιο τοξική ουσία της φύσης και για πάρα πολλά χρόνια η επιστημονική κοινότητα έλεγε ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσουμε ε, τους ποντικούς στον έλεγχο της τοξικότητας του μποτόξ. Επειδή το μποτόξ έχει ε, καλλιντική χρήση ε, τότε η ε, κοινή γνώμη έπεισε τους κατασκευαστές ε, του Μποτόξ στις Ηνωμένε Πολιτείες ότι μπορεί να πέσουν, να μειωθούν τα κέρδη τους. Και τότε ξαφνικά η βιομηχανία όταν πίστηκε βρήκε μια νέα μέθοδο που βασίζεται στη χρήση των ανθρώπινων κυτάρων για την πιο τοξική ουσία της φύσης. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι η επιστήμη. Το θέμα είναι να κυκλοφορήσει ένα πολύ περίπλοκο μήνυμα το οποίο σήμερα δεν πετύχαμε με τα δεκάλεπτα. Απαιτείται να υπάρξει μια σοβαρή επιστημονική συζήτηση την οποία θα κερδίσουμε νομίζω. Αυτή τη στιγμή στο κοινό συνειδητοποιήσει ότι τα πειράματα στα ζώα δεν είναι ένα αναγκαίο κακό που μας πουλάνε εδώ και χρόνια. Δεν είναι αναγκαίο πλέον, είναι μόνο κακό πράγμα. Η τεχνολογία υπάρχει, η κοινή γνώμη δεν θα αποδεχθεί πλέον το κακό και θα το απομακρύνει. ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę. Σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι ολοκληρώνεται ο τρίτος γύρος παρουσιάσεων και παρακαλώ τον κύριο Κμίνο, τα μήνα να πάρει τον λόγο για να καταλήξουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η ευρύτατη συζήτηση που δεν μπόρεσε να διευκρινίσει όλα τα επιστημονικά ζητήματα όπως υπόθηκε από τις προσθέσεις πλευρές, έχει νομίζω όμως φωτίσει κάποια στοιχεία πολύ σαφή και συγκεκριμένα προβλήματα. Εάν, όπως λίγο πολύ προκύπτει από κάθε πλευρά, δεχθούμε ότι δεν είναι προγνωστικοί οι πειραματισμοί του στα ζώα και εάν πούμε ότι απαιτείται από τη συνθήκη τη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η εγγύηση για την προστασία της ε, υγείας των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφού δεν υπάρχει τίποτα, χειρό, τίποτα καλύτερο πρέπει να χρησιμοποιούμε μια μέθοδο εσφαλμένη. Γιατί η μέθοδο εσφαλμένη παραμένει εσφαλμένη. Δεν είναι ότι ε, ελλείψη εναλλακτικών μετατρέπεται σε ορθή μέθοδο. Πρέπει όμως να βρούμε τρόπους, όρους με τους οποίους να μπορεί να αντικατασταθεί αυτή η εσφαλμένη μέθοδος. Ζητείται λοιπόν η, κατα η κατάργηση της οδηγίας, αυτή καθ' αυτή και τίποτε περισσότερο. Αυτό δεν αρκεί όμως. Υπάρχουν επιχειρήματα που λένε α, πρέπει με τις συνθήκες που ισχύουν τώρα να δούμε αν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η οδηγία έστω όπως έχει. Μα δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για την ευζοία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα για να μην υπάρχουν ζώα, πειραματόζωα πλέον. Οι επιλογές μας είναι πάνω απ' όλα όμως επιστημονικές όχι τόσο της ευζοβίας των ζώων. Δηλαδή πρέπει η πρώτη μας πρωταρχική μας υποχρέωση είναι να εξασφαλίσουμε την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του καταναλωτή και βέβαια του περιβάλλοντος. Άρα θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο αυτό όχι αύριο, εξάπαντος, είναι πολλά τα τεχνικά προβλήματα, το ξέρουμε, αλλά έχοντας δει ότι όταν ορίζουμε, από την εμπειρία μας, ότι όταν ορίζουμε προθεσμίες όπως ο Horizon 2020 κτλ. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι θέλουμε λίγο πολύ εκείνη την εποχή να έχουμε μια πραγματική πρόοδο η οποία να εξασφαλίζει την ε, διαφυγή από την αναγκαιότητα να γίνονται πειράματα σε ζώα. Άρα λοιπόν είναι πολύ αντιφατικό να έχουμε μια οδηγία η οποία από τη μια μεριά μας λέει ότι ο στόχος είναι η εν τέλει αντικατάσταση των πειραμάτων σε ζώα, ενώ από την άλλη λέει ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η χρησμή πειραματοζώων για την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Τέτοιου είδου εσωτερική αντίφαση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Και γι' αυτό εμεί ζητούμε να βγει αυτή η φράση και να σταματήσει αδίποτε αναφορά στην αναγκαιότητα των πειραμάτων σε ζώα. Αλλά βεβαίω και θα πρέπει μέσα σε ορθολογικού ρυθμούς να προχωρήσουμε σε μια αντικατάσταση με άλλε μεθόδου. Ε, λέγεται ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν οι μέθοδοι αντικαταστήσεις τα κάθε τι. Έστω. Ναι, αλλά άμα δεν δοθούν τα οικονομικά μέσα και η δυνατότητα τη έρευνα που θα απαιτηθεί, προφανώ και δεν πρόκειται να λύσουν τίποτα. Αν δεν θέλουμε κανένα αποτέλεσμα, αρκεί να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να προσφέρει πλέον το αποτέλεσμα αυτό που δεν θα έχουμε τα τεχνικά εργαλεία για να αντικαταστήσουμε τα πειράματα σε ζώα. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που θέλουμε να βρούμε μία μέθοδο, όχι τόσο αντικατάσταση ω προς την αποτελεσματικότητα, αλλά ω προς τη χρήση των ζώων και πιο αποτελεσματικός προς τη χρήση των ζώων, πρέπει αυτό να επιδιώκεται. Είναι μια επιλογή πολιτική, μια βούληση να διαθέσουμε τα απαραίτητα μέσα και για να απαντήσω και σε μια σειρά από επιφυλάξεις που ακούστηκαν, μέσα σε δύο χρόνια μπορούμε να προβλέψουμε να οργανώσουν οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια μεγάλη διάσκεψη ώστε με τρόπο αποτελεσματικό, ξεκάθαρο, επιστημονικό να αντιπαρατεθούν όλες οι απόψεις για να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα. Εμείς ετοιμάσαμε ένα φάκελο που ε, περιέχει ευρύτατη βιβλιογραφία που επιχειρηματολογεί υπέρ των θέσεών μας, τη διαθέση όλων των βουλευτών, αλλά δια του διαδικτύου θα είναι προσβάσιμο στους πάντες, χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, άλλωστε είναι πολύ εύκολο να βρεθεί, να, να αναζητήσει κανείς και να βρει όλα αυτά τα στοιχεία τα επιστημονικά. Α, θέλουμε όμως να δοθεί η δυνατότητα για μια σοβαρή αντιπαράθεση των θέσεων με χρόνους επαρκής, γιατί όταν είναι περιορισμένος ο χρόνος απλουστεύουμε, υπεραπλουστεύουμε, φτάνουμε στο είμαι υπέρ, είμαι κατά. Δεν αρκεί αυτό. Αυτό εμεί προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δοθεί επαρκή χρόνο σε συζήτηση. Και προτείνουμε επίση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν λέγεται ότι υπάρχουν πραγματικέ μέθοδοι αντικατάσταση που δεν θέλουν να πετούν, δηλαδή χρήση ζώων, αυτέ να, ε, ε, να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Το όντι το προβλέπει το άρθρο 4, αλλά για να κοιτάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο έχει τηρηθεί αυτό το άρθρο και όχι μόνο αυτό, και άλλε διατάξει, γιατί δεν χρειάζεται να κοιτάμε μόνο τι διατάξει σχετικέ με την προστασία των ζώων. Για να δούμε λίγο τι διατάξει και την εφαρμογή ε, σε σχέση με τις χημικές ουσίες. Το REACH, τα, τα βιοκτώνα, τα, ζω, τα ζυζανιοκτώνα, τη χρήση πρόσθετων στις, ε, στα τρόφιμα. Λίγο πολύ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι καλύτερο είναι πάντα να χρησιμοποιούνται τα ζώα. Δεν ε, αρκεί να υπάρχει αυτή η εγγύηση ότι κάθε φορά που έχει επιβεβαιωθεί μια εναλλακτική μέθοδος αυτή αποκλειστικά θα χρησιμοποιείται. Στη δε επικύρωση, η επικύρωση θα πρέπει να γίνεται πράγματι με κατάλληλο τρόπο με χρηματοδότηση επαρκή, με δομή, δομές, υφιστάμενες δομές ευρωπαϊκές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και με οικονομικά και επιστημονικά μέσα και ανθρώπινους πόρους και επαρκή. Η μέθοδος αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η μέθοδος που θα μας λέει εάν υπάρχει ένα σύστημα εναλλακτικό αυτού του πειράματος στα ζώα. Φαρμακολογικό είναι, τοξικολογικό είναι, έχουμε μία σειρά από δεδομένα για τις συνέπειες στον άνθρωπο, όλων αυτών που δυστυχώς έχει ε, περάσει ο άνθρωπος, γιατί ό,τι και να κάνουμε και όσα πειράματα και αν καταργήσουμε στα ζώα, το πραγματικό πειραματόζωο θα είναι τελικά ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αλλά έχουμε αρκετά στοιχεία ώστε να λέμε ότι υπάρχει μία μέθοδος που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να περάσει πια στην κλινική δοκιμή στον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να έχουμε μια ετήσια έκθεση, για να είμαστε και διαφανείς, ως προς την εφαρμογή και επιλογή των εναλλακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, δεχόμαστε τις διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή μας πάντα. Πάντα υπάρχουν καλές προθέσεις, αυτό είναι δεδομένο ότι η ποικιλία των θέσεων υπαγορεύεται από τις καλές προθέσεις. Υπάρχει μια σειρά από προτάσεις για την προστασία της ευημερίας των ζώων και της ευζοίας των ζώων. Δεν πρέπει όμω να λησμονούμε και τα όρια της επιστήμης. Η πρόταση για τη οργάνωση μιας μεγάλης διάσκεψης στο θέμα αυτό είναι μια πρόταση λογική. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το συμπέρασμα, το κύριο συμπέρασμα της σημερινής μας ακρόασης. Το μήνυμα που θα διαβάσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στις περιβαλλοντικές, στις κοινοβουλευτικές μας επιτροπές για το περιβάλλον, για τις αναφορές, οι οποίες ε, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούν να γίνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ του οργανωτέ τη πρωτοβουλία των πολιτών, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που μα αφύπνισε ω προ την ανάγκη να είμαστε σε επαγρύπνηση για το θέμα αυτό. Ε, είναι πια η ώρα να δώσουμε το λόγο σε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή αν προτιμάτε να περιμένουμε να καταλήξει σε απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοδότηση μπορεί να βρεθεί από τον το 2020. Ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμη για την υλοποίηση των ιδεών που ακούστηκαν στην ακρόασή μας. Ευχαριστώ τους πάντες και τις πάσες και πάνω απ' όλα τους 1 εκατομμύριο και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν στην πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ τους εργανωτές της πρωτοβουλίας για όλες τους τις προσπάθειες και κυρίως έτσι το πέρας της συνδυασίας μας. Σας εύχομαι. Καλό απόγευμα, καλή βραδιά και είστε επανειδήν για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα στο εγγύς μέλλον.